Thank you. Can we uh, start? We've already had a break for um, before. Είχαμε λοιπόν διακόψει, περιμένοντας την κυρία Όμεν. Σας παρακαλώ, καθίστε γρήγορα γρήγορα κυρία Όμεν. Πρέπει μέχρι τις 10 παρα 5 να έχουμε ολοκληρώσει και δεν πρόκειται να υπερβούμε αυτό το χρόνο. Άρα όσοι δεν έχουν μιλήσει ίσως έχουμε πρόβλημα. Επαναλαμβάνω, πρέπει ακριβώς 10 παρα 5 να έχουμε τελειώσει. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Όμεν Ρόιμεν να μας ε, μιλήσει για την έκθεσή της. Ζητώ συγγνώμη. Είχαμε τον Ολλανδό Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στο γραφείο μας. Και λυπάμαι που άργησα και δεν μπόρεσα να είμαι ακριβώς στις 9 εδώ. Ο συντονιστή, ο κ. Στράβο, ήταν πολύ πιο ε, γρήγορο στην επεξεργασία των δικών του θεμάτων από ό,τι νόμιζαν. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι συνεργαστήκαμε εξαιρετικά με τους σκιώδεις εισηγητές και από την αρχή δεσμεύτηκα έτσι ώστε να πετύχουμε μια συμφωνία εδώ στην Επιτροπή. Γιατί θεωρώ ότι ο προϋπολογισμός για τα συνταξιοδοτικά ταμεία είναι πολύ σημαντικός και για τώρα αλλά και για αργότερα. Η Πράσινη Βίβλος έχει σαν σκοπό να βρούμε ένα σύστημα ασφαλές, ένα σύστημα βιώσιμο, το οποίο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών. Συνεργαστήκαμε με έναν πάρα πολύ διαφανή τρόπο. Κάθε φορά δηλαδή που υπήρχαν τροπολογίες, κάθε φορά που εξέτασα τροπολογίες, προσπάθησα να υποβάλω συμβιβαστικά κείμενα τα συμβιβαστικά κείμενα αυτά. Φυσικά τα συζήτησα κάθε φορά και με τους κοιόδες εισηγητές, το οποίο ευχαριστώ ιδιαίτερα. Κύριε Πρόεδρε, το αποτέλεσμα αυτών των συζητήσεων είναι οι συμβιβαστικές τροπολογίες που βλέπετε ε, μπροστά σας, στο φακελό σας. Υπάρχουν δύο σημεία, μάλλον τρία σημεία, στα οποία μπορούμε να πούμε ότι συνεχίζουν να υπάρχουν δυσκολίες. Πρώτο σημείο. σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης, μέσα στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι συντάξεις. Αυτό που θα θέλαμε να ξέρουμε είναι κατά πόσο έχουν ληφθεί συντάξεις υπόψη στο πακέτο αυτό. Γι' αυτό και την προηγούμενη εβδομάδα, ακριβώς επειδή δεν μπορέσαμε να συμφωνήσουμε 100% ζητήσαμε από τον εκπρόσωπο της ΕΚΦΙΝ στην Επιτροπή να μας δώσει κάποιες εξηγήσεις. Σήμερα ξέρουμε ότι όντως οι σε ελήφθησαν υπόψη στο Σύμφωνο Ανάπτυξης και Σταθερότητας. Αυτό που δεν ξέρουμε ακόμα είναι πώς ακριβώς. Και βεβαίως αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Και δεν νομίζω ότι διαφέρουν εδώ οι απόψεις μου από αυτές των άλλων. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που υπάρχει δέσμευση για τον πρώτο πυλώνα, αυτή η υποχρέωση, αυτή η δέσμευση έχει συνέπειες. Αυτό μου φαίνεται ότι είναι σαφές. Συνέπειες επί της ανάπτυξης και της σταθερότητας και τα κράτη-μέλη κάνουν εξοικονομήσεις για μια συμπληρωματική, παραδείγματο χάρη, πρόβλεψη ε, για συντάξεις αυξάνονται την ίδια ώρα και οι δαπάνες των κρατών μελών αυξάνεται και το χρέος των κρατών μελών. Εμείς θεωρούμε ότι εδώ πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για κάθε τέτοιου είδους ε, εξοικονόμηση που κάνουν τα κράτη-μέλη. Και αυτό το αναφέρουμε στην παράγραφο 5. Κυρία Πρόεδρε, προσπάθησα να ικανοποιήσω όλες τις ε, πλευρές. Διαπιστώνω βεβαίως ότι υπάρχει συμβαστική πρόταση ε και σαφώς εδώ θα πρέπει να συμπληρωθεί το κείμενο. Η Οικονομική Επιτροπή μας έχει υποβάλει τρεις παραγράφους. Ίσως είναι λίγο πολύ αυτή η προσθήκη εδώ, τρεις επιπλέον παράγραφοι. Παρ' όλα αυτά δεν βλέπω πώς μπορούμε να μην τους συμπεριλάβουμε, να μην συμπεριλάβουμε αυτές τις προτάσεις. Πιστεύω ότι η σοσιαλιστική ομάδα θα υποστηρίξει. Εγώ προσωπικά δεν είμαι αντίθετη με την ε, πρόταση αυτή της τρεις επιπλέον παράγραφος. Τώρα, όσον αφορά τους πυλώνες, η... το σημείο εκκίνησης της έκθεσης αυτής είναι ο πρώτος πυλώνας, δηλαδή το σύστημα που βασίζεται στην αλληλεγγύη, το σύστημα που χρηματοδοτείται από από τα κράτη. Αυτός είναι ο πρώτος και βασικός πυλώνας. Βεβαίως εξαιτίας της γύρανσης του πληθυσμού όλο και λιγότερο νέοι εργαζόμενοι συνεισφέρουν στο σύστημα. Αυξάνεται ο αριθμός των ηλικιωμένων στις κοινωνίες μας, αυξάνεται ο αριθμός των ατόμων που δεν μπορούν να συνεισφέρουν. Το δεύτερο λοιπόν σημείο είναι ο δεύτερος πυλώνας ο δεύτερος πυλώνας που συνεχίζει να απορρέει από την εργασιακή σχέση μεταξύ ενός εργοδότη και ενός εργαζόμενου. Κάποια χρήματα χρηματοδοτούν την λεγόμενη συμπληρωματική σύνταξη. Στη Γερμανία, παραδείγματο χάρη, έχουμε ένα πολύ ε, σαφές ε, μοντέλο αυτής της συμπληρωματικής ε, χρηματοδότησης. Σε πολλές χώρες βεβαίως υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι κερδίζουν αρκετά έτσι ώστε να εξοικονομήσουν κάποια ποσά. Αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι ένα γενικευμένο σύστημα σε καμία περίπτωση. Τρίτο σημείο κυρία Πρόεδρε, για το οποίο πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει ακόμα καμία συμφωνία. Όπως ε, λέω στην έκθεση, η γύρανση του πληθυσμού είναι ένα γενικευμένο φαινόμενο. Ο αριθμός των ηλικιωμένων αυξάνεται και η αύξηση του προσδόκιμου ζωής βεβαίως είναι ένα φαινόμενο που χαρακτηρίζει όλες τις χώρες αλλά σε πολύ διαφορετικό βαθμό. Για τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, παραδείγματο χάρη, 68 ετών είναι το προσδόκιμο ηλικία. Στην Ολλανδία, 79 για τους άντρες. Ανάλογα λοιπόν με τη χώρα που, ζου, που ζει κάποιος, υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Γι' αυτό και παρατηρούμε πολύ σημαντική διαφορά και στις προτάσεις των συναδέλφων. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν αυτοί που λένε ότι δεν θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας αυτές τις σημαντικές διαφορές και ότι θα πρέπει να συνεχίσουν να εργάζονται οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι όσο είναι σε θέση να εργαστούν. Να υπάρχει δηλαδή μεγάλη ευελιξία και το όριο συνταξιοδότησης να μην είναι πολύ νωρίς. Εγώ αυτό που είπα είναι ότι δεν είναι δυνατόν να πούμε ότι θα υπάρχει όριο συνταξιοδότησης για όλη την Ευρώπη. Αυτό δεν είναι δυνατόν. Είναι μια γερμανική πρόταση, η πρόταση της κυρίας Μέρκελ. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε με τους κοινωνικούς εταίρους, με όλους τους εργαζόμενους, πώς μπορούμε να κοιτάξουμε ανακράτος μέλος την ιδιαίτερη κατάσταση που επικρατεί στις χώρες. Νομίζω ότι η συνεισφορά των κοινωνικών εταίρων είναι καθοριστική στο σημείο αυτό και ελπίζω να με υποστηρίξουν οι σοσιαλιστές συνάδελφοι στην πρόταση που κάνω ε, στο κείμενό μου για το θέμα αυτό. Αναφέρομαι στο συμβιβαστικό κείμενο S, σίγμα, για την παράγραφο 18. Αυτά ήθελα να πω καταρχήν κυρία Πρόεδρε και πραγματικά ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να φτάσουμε μετά από την επεξεργασία σε μια καλή έκθεση, σε ένα καλό κείμενο το οποίο θα μπορέσουν να υποστήριξουν όλοι. Είμαι στη διάθεσή σας βεβαίως αν έχετε ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Τόμας όχι, Μαρι Χόπκιν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια που ο τρόπος με τον οποίο εργάστηκε τουλάχιστον κατ' εμέ διευκόλυνε το έργο και των σκιωδών ε, εισηγητών. Και την ευχαριστώ όπως και τους συνεργάτες μας. Έχω κάποια θέματα. Πρώτα απ' όλα σε ό,τι αφορά την συμβιβαστική ε, ΣΥ. Θα ήθελα μία επεξήγηση μιλάει για την ανάπτυξη διακλαδικών ή και εδαφικών ταμείων για να αυξηθεί η συμμετοχή των εργαζομένων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στα εξοδοτικά συστήματα. Τι θα πει ακριβώς το territorial funds, εδαφικά ταμεία και πώς αυτό θα αυξήσει την συμμετοχή, των, την εγγραφή των εργαζομένων στα ταμεία. Θέλω κάποια επεξήγηση σε αυτό. Δεύτερον, ε, στο, ε, σε ό,τι αφορά τη συμβιβαστική age πράγματι είναι πολύ σημαντικό ότι πρέπει να είναι επαρκής και οι συντάξεις ε, των γυναικών. Σε ό,τι αφορά τώρα τους τρεις πυλώνες ε, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Εγώ συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με την εισηγήτρια και η ομάδα μου θα στηρίξει τις τροπολογίες. Τώρα, σε ό,τι αφορά την συμβιβαστική ΆΗ, Στην πρώτη πρόταση λέγεται ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν θετικά κριτήρια τον υπολογισμό των συντάξεων των γυναικών. Εγώ θα έλεγα ότι η λέξη positive, θετικά, μάλλον πρέπει να διαγραφεί γιατί στην επόμενη πρόταση λέγεται ότι κατά τρόπο ώστε να είναι εγγυημένη οικονομική ανεξαρτησία και των ανδρών και των γυναικών. Νομίζω λοιπόν ότι περιτεύει η λέξη θετικά γιατί χαρακτηρίζει κατά κάποιο τρόπο την έκθεση και είναι και λίγο ύποπτος όρος θετικά κριτήρια. Όμως η λέξη αυτή δεν κάνει πιο σαφή τη διατύπωση, η οποία είναι ήδη με την φράση την επόμενη. Ίσως λοιπόν δημιουργηθούν κάποια ζητήματα. Τώρα, ηλικία συνταξιοδότησης και πάλι συμφωνώ δεν χρειάζεται να κάνουμε εναρμόνιση θα μπορούσε να συνδεθεί με το προσδόκιμο ζωή, Αυτό θα αποφασιστεί σε επίπεδο κρατών μελών κτλ. Το τελευταίο μου σχόλιο αφορά τι ε, τροπολογίε τη επιτροπή ΕΚΟΝ και το Σύμφωνο ανάπτυξη και Σταθερότητα. Όπως είπε και η συγγετρία, περιλαμβάνονται οι συντάξεις, αλλά είναι πολύ δύσκολο να δει κανεί και σε ποιο βαθμό και με ποιο τρόπο. Αυτό είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα για τα κράτη-μέλη. Αν δείτε την παράγραφο 9, για παράδειγμα, για την οίκον μιλάω, είναι σαφέστατο ότι θέλει να λαμβάνονται υπόψη μεταρρυθμίσεις των συνταξιοδοτικών συστημάτων στη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος και λέει έπειτα ότι φραστή θλίπτη λείπτη για το ότι ε, έχουν αλλάξει κάποια ε, κράτη-μέλη ε, τις διατάξεις τι με τις συντάξεις για να κάνουν κάποιες περικοπές. Εγώ προέρχομαι από μια χώρα που δεν είχαμε άλλη επιλογή Ουσιαστικά το, ΆΙ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ε, μας έδωσε και το Σύμφωνο Σταθερότητας, μας έδωσε αυτή την εντολή. Μας κατήφινε προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχει λοιπόν μια αντίφαση και νομίζω ότι είναι λίγο ατυχές που είναι το 2, το 9 και το 10 στην έκθεση, λόγω της αβεβαιότητας που υπάρχει. Αλλά η ομάδα μου παρόλα αυτά μάλλον θα μπορέσει να στηρίξει Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε, Μάριαν. Τόμας Μαν, τώρα και μετά κύριε Σάρι. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Πιστεύω ότι τις τελευταίες εβδομάδες η εργασία αυτή πραγματικά έφερε αποτελέσματα. Υπήρξε εξαιρετική συνεργασία, όχι μόνο με τους ε, σκιώδεις. Δεν ήταν εύκολο αυτό που έκανε η συγγήτρια μέχρι να φτάσουμε τελικά σε αυτές τις συμβαστικές προτάσεις. Πραγματικά ήταν πολύ καλή η συζήτηση που είχαμε, επικοδομητική. Είδαμε και τις προτάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, οι τροπολογίες οίκων δεν θα συμπεριληφθούν στην ψηφοφορία. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που συμπεριλαμβάνουν. Θεωρώ πολύ ουσιαστικό το ότι καταφέραμε να φτάσουμε σε κάποιες ε, συμβιβαστικές τροπολογίες με μεγάλη ε, στήριξη, γιατί διαπιστώνουμε, ε, κοιτώντας το θέμα αυτό, πόσο διαφορετικά είναι τα συστήματα, η πραγματικότητα στις διάφορες χώρες. Πόσο διαφορετικά είναι αυτά που έχουν πετύχει οι εργαζόμενοι και πόσο διαφορετική είναι η κατάσταση. Αυτό που έχει σημασία είναι να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε αυτές τις διαφορές με την συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και να δούμε πώς μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας τις ομοιότητες και τις διαφορές. Υπάρχουν κρατή-μέλη που έχουν παρόμοια συστήματα. Μιλήσαμε, παραδείγματος χάρη στη συμβαστική τροπολογία ΔΕΛΤΑ, για τα ελάχιστα επιτεύγματα και πρότυπα. Και βεβαίως εδώ αναφερόμαστε στην διασυνοριακή αν θέλετε, κίνηση των εργαζομένων εδώ πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να ε, προσπαθήσουμε να ρυθμίσουμε αυτή τη διασυνοριακή ε, κυκλοφορία των εργαζομένων, αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι εδώ να προσέξουμε ιδιαίτερα αυτό που ονομάζουμε minimum standards, τα ελάχιστα δηλαδή ε, πρότυπα και είναι πολύ σημαντικό όπως αναφέρουμε και στην πράσινη βίβλο και όταν βεβαίως φτάσουμε στην Λευκή Βίβλο της Επιτροπής. Είναι κάτι το οποίο έχει μεγάλη κυκλοφορία και πρέπει να δούμε ότι όπως φαίνεται εξάλλου όταν κοιτάξει κανείς τις τροπολογίες της ε, εικόν και ιδιαίτερα στο σημείο 50 ότι όλα αυτά τα διαφορετικά σημεία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται. Και νομίζω ότι αυτό είναι το καλό που πετύχαμε συμβαστικές τροπολογίες, ότι όλες αυτές οι διαφορές, διαφορετικές προσεγγίσεις έχουν ληφθεί υπόψη και ότι αυτό θα πρέπει να το συνεχίσουμε και στην περαιτέρω επεξεργασία και όταν φτάσουμε στη Λευκή Βίβλο ελπίζω οι διαφορές να έχουν μειωθεί. Ναι, ευελιξία, ναι, κινητικότητα, αλλά όταν μιλάμε για θέματα κοινωνικής πολιτικής θα πρέπει και οι κοινωνικοί εταίροι να μπορούν να συμμετάχουν πλήρως. Ο κύριος Σέρ, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα συνεχίσω εκεί που σταμάτησε ο Τόμας Μαν. Και εγώ θεωρώ ότι πραγματικά αυτή η πρώτη φάση της συζήτησης ε, δίρκεσε πολύ. Αναγκαστήκαμε να επεξεργαστούμε όλα αυτά τα θέματα μαζί για να μπορέσουμε να αναφερθούμε όσον αφορά την πράσινη βίβλο και τις πρώτες αυτές προτάσεις. Ήταν πολύ επικοδομητική η εργασία μας και ευχαριστώ ιδιαίτερα την συγγήτρια, την κυρία Ομεν Ρόιτεν και την εργασία της. Πολλές ε, προτάσεις από τις οποίες κατάφερε να δημιουργήσει ένα συμβιβαστικό κείμενο. Και αυτό δεν ήταν εύκολο. Βεβαίως δεν λέω ότι το κείμενο αυτό μπορεί να καλύψει όλες τις προτάσεις. Μία συμβιβαστική λύση δεν μπορεί να ικανοποιήσει όλες τις πλευρές, δεν μπορεί να καλύψει όλες τις ε, διεκδικήσεις και προτάσεις. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι εδώ πετύχαμε κάτι που είναι αρκετά ρεαλιστικό και βεβαίως οι διάφορες πολιτικές ομάδες, τα κράτη-μέλη, το Κοινοβούλιο θα δουν τι από αυτά μπορούν να λειτουργήσουν με ικανοποιητικό τρόπο. Στο ΕΛΚ μπορούμε να στηρίξουμε την συμβαστική αυτή πρόταση. Γι' αυτό και έχουμε αποσύρει τις περισσότερες από τις τροπολογίες μας για να μπορέσει να προχωρήσει αυτή η συμβαστική πρόταση. Όσον αφορά τις παρατηρήσεις της Μαρίας Νάρκιν, δεν λέω ότι διαφωνώ με αυτά που προτείνει η Οικονομική Επιτροπή. Αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι τα συστήματα είναι τελείως διαφορετικά στα κράτη-μέλη. Στην Ουγγαρία, παραδείγματος χάρη, εμείς μειώσαμε τα κρατικά ελλείμματα και την ίδια ώρα ξεκινήσαμε μια τεράστια μεταρρύθμιση. Δηλαδή, κάθε χρόνο 1,5 δις ευρώ βγαίνουν από τα συνταξιοδοτικά ταμεία Αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και από τις ουγγρικές επιχειρήσεις. Δημιουργήσαμε στη χώρα μου ένα σύστημα το οποίο προσπαθούμε να αλλάξουμε. Δεν ήταν σταθερό, δεν ήταν βιώσιμο. Και δεν μπορούμε να καταδικάσουμε αυτή τη στιγμή αυτήν την μεταρρύθμιση. Πρέπει να βρεθεί μια λύση. Πρέπει να βρεθεί μια λύση για χώρες όπως η Ιρλανδία, όπως η Ουγγαρία που προσπαθούν να μεταρρυθμίσουν τα συστήματά τους και αυτό είναι πάρα πολύ επίπονο. Ακριβώς γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι δεν πρέπει να αγνοούμε τις τεράστιες διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των συνταξιοδοτικών συστημάτων. Υπάρχει η Ιρλανδία, υπάρχουν και άλλα μοντέλα και πρέπει να δείξουμε ανοχή, να καταλάβουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κάποιες χώρες. Το θέμα των συντάξεων είναι εξαιρετικά σημαντικό για όλους μας. Και εμείς σε 10-15 χρόνια θα θέλαμε να έχουμε μια σύνταξη που να μας καλύπτει. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθούν αποδεκτές λύσεις. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν την Ρία και νομίζω ότι μπορούμε να δεχτούμε την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Δεν ήταν προφανές να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια που ξεκίνησε εδώ και κάποιες εβδομάδες σε σχέση με το σχέδιο έκθεσης. Ήταν ένα πολύπλοκο εγχείρημα, υπήρχαν διάφορες ευαισθησίες και μάλιστα και εντός ε, των πολιτικών ομάδων. Θα ήθελα να χαιρετήσω και να υπογραμμίσω την καλή δουλειά, τη σημαντική δουλειά και τις διαπραγματεύσεις που έφερε σε πέραση η Ρία. Θέλοντας να δώσει στο τελικό κείμενο, μια προβολή, ε, μια συνοχή και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό και αν θέλουμε να είμαστε όλοι μας αξιόπιστοι προς τα έξω και αν θέλουμε η έκθεση αυτή να επηρεάσει και το έργο του Επιτρόπου. Γιατί νομίζω ότι και αυτός είναι ένας από τους στόχους μας. Τώρα, σε σχέση με την πρόοδο των εργασιών μας, θα ήθελα να πω ότι είναι σε πολλά μέτωπα η πρόοδος αυτή. Θα ήθελα να τονίσω κάποια στοιχεία. Πρώτα απ' όλα, η θέση που δίνεται στους διάφορους πυλώνες ε, ξεκάθαρα ε, βέβαια στις συμβαστικές προτάσεις και όχι τόσο στην έκθεση τονίζει τη σημασία του πρώτου πυλώνα η μεγάλη σημασία που έχει είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της αλληλεγγύης αλλά και της ασφάλειας της χρηματοδότησης των συντάξεων αυτό νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό στοιχείο τώρα σε ό,τι αφορά το δεύτερο πυλώνα που αποτελεί μια πραγματικότητα λίγο, λιγότερο περισσότερο υπαρκτή στα διάφορα κράτη μελη γιατί νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε ενίσχυση του ρόλου του πυλώνα αυτού, αλλά σε συνεννόηση με τους κοινωνικούς εταίρους ε, που είναι οι πρωταρχικοί φορείς, όπως ε, αυτό μεταφράζεται και στις συμβιβαστικές προτάσεις. Είναι ένα στοιχείο που θέλω να το τονίσω. Τρίτος τώρα πυλώνας. Πρέπει να αναφερθεί, πρέπει να αναφερθεί όμως να διακριθεί αν θέλετε από τους δύο προηγούμενους δεν είναι η βάση για τη σύνταξη αλλά όπως αναφέρεται και στις ε, συμβιβαστικέ τροπολογίες Για όσους έχουν τις δυνατότητες για όσους έχουν τα μέσα, μπορεί να αποτελέσει μια συμπληρωματική πηγή σύνταξη. Αυτό δεν μπορούμε να το αρνηθούμε, αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να ε, είναι και ένα θεμελιώδη πυλώνα. Αυτό είναι ένα πρώτο στοιχείο σε ό,τι αφορά τη θέση των πυλώνων. Ένα άλλο σχόλιο που θέλω να κάνω έχει να κάνει με την παράγραφο 5. Παράγραφος 5 είναι μια δύσκολη παράγραφος. Αποτέλεσε αντικείμενο πολλών συνεδριάσεων και συζητήσεων. Και στην τελευταία διατύπωση που έχω εδώ, η συμβαστική πρόταση μου φαίνεται αποδεκτή. Μου φαίνεται αποδεκτή. Παρόλα αυτά, θέλω να προσθέσω ένα στοιχείο. Η προσθήκη της παραγράφου που προέρχεται από την Επιτροπή ΕΚΟΝ. Δεν ξέρω κατά πόσον αυτό συνεισφέρει στο να έχουμε μεγαλύτερη προβολή. Υπάρχει κατανομή των αρμοδιοτήτων των διαφόρων επιτροπών, αλλά έχω την εντύπωση ότι παράγραφος 5, συμβαστική ε, η διατύπωσή της ε, νομίζω αρκούσε και δεν θα προσθέσει κάτι παραπάνω το κομμάτι που έχει να κάνει με την ΕΚΟ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη φορητότητα, και αυτό είναι λίγο δύσκολο γιατί υπάρχουν ιδιαιτερότητε που πρέπει να γίνουν σεβαστέ. Ιδιαιτερότητε σε κάθε χώρα. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Νομίζω συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει να ενισχυθεί ο διασυνοριακό χαρακτήρα τη ε, αγορά απασχόληση, αλλά από την άλλη πλευρά δεν θα πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο τα όσα ήδη υπάρχουν σε κάποιε χώρε. Άρα νομίζω ε, ότι πρέπει να υπάρξει επιδίωξη συμφιλίωσης των δύο αυτών πτυχών στη διατύπωση της έκθεσης και των συμβαστικών τροπολογιών. Τώρα, ηλικία συνταξιοδότησης. Για την ηλικία συνταξιοδότησης. Εγώ πάντα εξέφρασα τις ε, αμφιβολίες μου για το θέμα αυτό. Πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα όχι στην νομικά επιβαλόμενη ηλικία, αλλά στην ουσιαστική ηλικία συνταξιοδότησης. Και όταν συνδέουμε την ε, ηλικία συνταξιοδότησης στο προσδόκιμο επιβίωσης, αυτό δημιουργεί πολλές επιφυλάξεις, τουλάχιστον μέσα στη δική μου πολιτική ομάδα. Αλλά πιστεύω ότι ο τρόπος με τον οποίο έχουν διατυπωθεί τα πράγματα στη συμβαστική τροπολογία, όπου δεν υπάρχει αυτή η αυτόματη σύνδεση μεταξύ προσδόκιμου επιβίωσης και ηλικία συνταξιοδότησης αναφέρεται το ότι η κάθε χώρα θα πρέπει να προβεί σε προβληματισμό σε σχέση με τις καταστάσεις που έχει να αντιμετωπίσει όπου θα πρέπει να υπάρξει σημαντικός ρόλος των κοινωνικών εταίρων. Νομίζω ότι με αυτή την προβληματική θα μπορούσαμε να ανοίξουμε ένα γενικότερο διάλογο Σε κάποιες φορές υπάρχει αυτή η συζήτηση για τη σύνδεση των δύο αυτών στοιχείων, αλλά το να μην είναι αυτόματη αυτή η σύνδεση και να βρίσκεται στο, στο πλαίσιο νομίζω ότι θα είναι θετικό, ότι θα είναι πρόοδο σε σχέση με αυτά τα οποία επιζητούμε. Αυτές είναι λοιπόν οι λίγες σκέψεις μου σε σχέση με το περιεχόμενο των συμβιβαστικών αυτών τροπολογιών. Και όπως σας έλεγα, οι τροπολογίες των διαφορών ομάδων απηχούν διαφορετικές ευαισθησίες. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να ζητήσω από την, προσωπική μου, από την πολιτική μου ομάδα να υποστηρίξει αυτές τις συμβιβαστικές λύσεις και να μην υποστηρίξει τις τροπολογίες που μπορεί να είναι καλές επί της ουσίας, αλλά οι οποίες θα ανατρέψουν τις συμβιβαστικές λύσεις. Γιατί η συμβιβαστική λύση απαιτεί να δούνε και λαβήν, αλής βερίς. Και επομένως πολλές φορές ξεπερνούν τις επιθυμίες αυτών που συμβάλλουν σε αυτή τη συμβαστική τροπολογία. Δεν πρέπει να ανατρέψουμε λοιπόν τις συμβαστικές λύσεις. Ίσως μπορούν να αποσυρθούν κάποιες τροπολογίες. Εγώ θα αποσύρω και κάποιες τροπολογίες δικές μου. Δεν μπορώ φυσικά να δεσμευτώ εξ ονόματος όλων των συναδελφών της πολιτικής μου ομάδας, αλλά δεν πρέπει να έχουμε τροπολογίες οι οποίες θα θέσουν ένα αμφιβόλο τις συμβαστικές λύσεις. <clears throat> Υπάρχουν βέβαια και κάποιες τροπολογίες πιο περιθωριακού χαρακτήρα, αν θέλετε, που δεν εμποδίσουν τις ε, συμβαστικέ τροπολογίε να ευδοκιμήσουν και θα υποστηριχθούν από τη δική μα πολιτική ομάδα. Αυτή είναι η σκέψη λοιπόν τη ομάδα μα. Ευχαριστώ. Μένουμε από χρόνο σιγά σιγά. Θα ήθελα να παρακαλέσω τους υπόλοιπου ομιλητές να είναι σχετικά σύντιμοι. Κορνέλσεν, Κύριε Κορνέλσεν. Θα κάνω τι μπορώ. Έχω μεγάλο σεβασμό για τον εισηγητή, για την εισηγητρία, συγγνώμη. Νομίζω ότι έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά <clears throat> με τις συμβαστικές τροπολογίες σε αυτό το πολύ δύσκολο θέμα και παρόλα αυτά κατάφερε να διατηρήσει κάποιο περιεχόμενο στην έκθεση αυτή. Δύο πράγματα νομίζω ότι είναι παράδοξα ή λυπηρά αν θέλετε. Υπογραμμίζεται σε κάθε δυνατό σημείο η επικουρικότητα. Σωστό είναι αυτό αν τα κράτη-μέλη μπορούν να μεταρρυθμίσουν τα συνταξιδοτικά του συστήματα με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι και οικονομικά εύρωστα και συγχρόνως εμποδίσουν την ένδια σε μεγάλη ηλικία, θα πρέπει να έχουν την ελευθερία επιλογής του τρόπου με τον οποίο θα φέρουν σε πέρα αυτή την μεταρρύθμιση. Αυτό αφορά τα συστήματα με πολλούς πυλώνες, αλλά και το θέμα της ηλικίας συνταξιοδότησης. Αλλά όσο προσεκτικά και να είναι διατυπωμένο το σημείο αυτό, μία από τις συμβαστικές τροπολογίες <clears throat> προωθεί τη σύνδεση μεταξύ ηλικία συνταξιοδότηση και προσδοκίμου επιβίωση. Αυτό καταπατά κάπου την έννοια της επικουρικότητας. Εγώ πιστεύω ότι για το θέμα της βιωσιμότητας των συντάξεων μπορούμε να τις κάνουμε τα, βι... τα συνταξιοδοτικά ταμεία βιώσιμα, αλλά με το κόστος μεγάλης ένδυας στην ε, τρίτη ηλικία. Δεν είναι αυτό που θέλουμε. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι επαρκές <clears throat> να εμποδίσουμε μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα θέσουν σε κίνδυνο την βιωσιμότητα των ταμείων. Πρέπει να δούμε και την άλλη πτυγή. Αλλά παρόλα αυτά, εμείς ε, καλοδεχόμαστε αυτήν την έκθεση και ευχαριστούμε τη Ρία για το έργο της. Η Φιγκερέντου έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι φανερό ότι σε μια τέτοια έκθεση είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο της εισηγήτριας γιατί έχει να αντιμετωπίσει μια πολυπληθώρα προτάσεων από τις διάφορες πολιτικές ομάδες. Σε σχέση με τον τελικό απολογισμό των προτάσεων και των συμβιβαστικών λύσεων που επέτυχε η εισηγήτρια, είναι γεγονός ότι σε πολλέ περιπτώσεις οι βασικέ λύσει έχουν καταφέρει να βελτιώσουν το βασικό έγγραφο τη Κομισιόν και κάποιες από αυτές τι τροπολογίε θα μπορούσαμε εμεί να τι δεχτούμε, αλλά είναι πολλές αυτές τις οποίες δεν μπορούμε να δεχτούμε γιατί έχουμε μια διαφορετική άποψη. Για μας υπάρχουν τρία ουσιώδη θέματα τα οποία θέλω να υπογραμμίσω. Καταρχήν, ο πρώτος πυλών, ο οποίος πρέπει να είναι ένα βασικό στοιχείο της μεταρρύθμισης της, ε, του, των Ταμείων Συνταξιοδότησης που πρέπει να είναι δημόσια, πρέπει να είναι αλληλέγγυα και θα πρέπει να προωθούν και την απασχόληση. Ξέρουμε <clears throat> ότι πολλά από τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν είναι και αποτέλεσμα της μεγάλης ανεργίας. Αν οι νέε γενναίες δεν είχαν ανεργία μεταξύ 20 και 40% σε ορισμένες χώρες, πάνω από 40% ανεργία των νέων, αυτό δεν θα ήταν αισθητό στα συστήματα συνταξιοδότησης, τα οποία έχουν ήδη προβλήματα ως εκ του τούτου. Επομένως, η πρώτη γραμμή άμυνας των δημοσίων συστημάτων συνταξιοδότησης είναι ακριβώς το να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης για τις νέες γενιές. Αυτό είναι βασικό και ουσιαστικό. Και θα πρέπει να τονίσουμε πάρα πολύ την ε, επιδίωξη αυτή. Εμεί φυσικά δεν θέλουμε να υπάρχει ηλικία συνταξιοδότηση που να είναι ίδια σε όλα τα κράτη, γιατί υπάρχουν διαφορετικές παραδόσεις και συνθήκες, αλλά δεν θέλουμε να υπάρχει και άμεση σύνδεση μεταξύ προσδοκίου επιβίωση και ηλικία συνταξιοδότηση. Αυτό προσπαθήσαν να το κάνουν στην Πορτογαλία και αυτή τη στιγμή ήδη χάνουν πάρα πολλοί συνταξιούχοι από τις μεταρρυθμίσεις. Και οι μελέτες Περιμένουμε ότι θα είναι πολύ περισσότεροι αυτοί οι οποίοι θα συνταξιοδοτηθούν τα επόμενα χρόνια. Επομένω αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα. Εμείς λοιπόν μετά από την εμπειρία της Πορτογαλίας είμαστε εναντίον μιας τέτοια σύνδεσης. Και το τελευταίο σημείο το οποίο θέλω να θίξω είναι ότι για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την ένδια, ένα από τα βασικά εργαλεία που έχουμε στην διάθεσή μας είναι να υπάρχουν ελάχιστες συντάξεις οι οποίες να εξασφαλίσουν μια ζωή με ε, αξιοπρέπεια στα άτομα τα οποία έχουν συνταξιοδοτηθεί. Δυστυχώ οι στατιστικές το καταδεικνύουν σε πολλά κρατημέλη και φυσικά και στη δική μου χώρα. Ένα μεγάλο μέρο των συνταξιοδοτουμένων, ιδίω των γυναικών, ζουν σε καταστάσει ένδυα, γιατί οι ελάχιστε συντάξεις δεν τους επιτρέπουν να ζήσουν σε ένα επίπεδο αξιοπρεπές. Οι ελάχιστες συντάξεις στη χώρα μου είναι μικρότερες και από το ίμιση του κατοφλίου ένδυας. Η... Η... Η ελάχιστο... Ο ελάχιστος μισθός στην Πορτογαλία είναι 485 ευρώ. Αλλά έχουμε στην Πορτογαλία συντάξεις που είναι της τάξης των 200 ευρώ το μήνα μονάχα και ιδίω για τι γυναίκε. Και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα μια κατάσταση έντονη ένδυας. Για αυτό το λόγο θεωρώ ότι αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν λαμβάνεται επαρκώ υπόψη στην έκθεση της κυρία Όμεν Ρόιντ και νομίζω ότι είναι και ένα συζήτημα το οποίο είναι κεφαλαιόδες για να αντιμετωπίσουμε την ε, ένδυα στα κράτη-μέλη. Αυτοί είναι οι κύριοι λόγοι για του οποίου μα ε, οδηγούν πρώτον το να μην αποσύρουμε τις δικές μας τροπολογίες και δεύτερον να επιμείνουμε ότι πρέπει να υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση σε σχέση με το θέμα αυτό, γιατί πρέπει να πριτανεύσει η ανάγκη του αγώνα κατά της ε, ένδυας, να υποστηριχθεί η περισσότερη απασχόληση για τους νέους και να υπάρχει δυνατότητα μιας αξιοπρεπούς ε, ζωής μετά τη συνταξιοδότηση και ιδίως ίσων δικαιωμάτων για άνδρες και γυναίκες. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομη. Πρώτα απ' όλα, κύριε Γκέρλινγκ, θέλω να ευχαριστήσω και εγώ την εισηγήτρια για το ανοιχτό πνεύμα με το οποίο εργάστηκε. Η μόνη μου, έτσι, το μόνο μου παράπονο ότι ακόμα δεν ε, μπορώ να προφέρω ακόμη σωστά το όνομα της κυρίας Συγήτης. Τέλος πάντων, το θέμα της επικουρικότητας είναι κάτι που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Επίσης, ε, θέλουμε να υπάρχει ένα επαρκές εισόδημα και να υπάρχουν τα επαρκή κονδύλια. Αυτό είναι ένα εθνικό προνόμιο που βασίζεται στις επιλογές ε, στο εθνικό επίπεδο. Παρ' όλα αυτά, προσπαθούμε να καταλήξουμε σε συμβαστικές λύσεις επί των οποίων να μπορούμε και εμείς να συμφωνήσουμε και θέλω να αναφέρω τρεις τομείς επί των οποίων δεν είμαστε σίγουροι αν μπορούμε να στηρίξουμε ή όχι. Πρώτον, Συμβεβαστική I. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Χάρκιν που λέει να παλύψουμε τη λέξη positive, θετικά. Έτσι θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε. Σε ό,τι αφορά τώρα τη συμβαστική J και πάλι χαίρομαι που λέμε για τα επαρκή κατώτατα επίπεδα που πρέπει να θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά και πάλι γίνεται λόγο για κριτήρια για τη θέσπιση κατωτάτων επίπεδων σε επίπεδο κρατών μελών. Και το πρέπει να καθοριστεί από την Κομισιόν. Εγώ δεν βλέπω λόγο για κάτι τέτοιο, αυτό δεν μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Τέλο, β, λατινικό, για την κατάρτιση νέων δικτών. σω φαίνεται κάτι όχι τόσο σημαντικό αλλά ε, είχαμε συμφωνήσει το 2001 δείκτες και δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτοί οι δείκτες είναι ανεπαρκείς και πρέπει να αλλάξουν. Και δεν ξέρω για ποιο λόγο τελικά θέλουμε μια συμβιβαστική πρόταση η οποία να λέει για νέους δείκτες. Άρα ούτε εδώ είμαστε ικανοποιημένοι. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, πριν δώσω το λόγο και πάλι στην κυρία Ρόιτεν για την συμβιβαστική Q και την τροπολογία τη δική μου 233. Θέλω να πω το εξή. Πολλοί από εσά νομίζω κάντε, ε, κάπως συγχύσατε λίγο τα πράγματα. Εγώ στην 233 έλεγα αν μπορούμε να δούμε τη σκοπιμότητα θέλαμε να υπάρχει η, κατά το, η νόμα προβλεπόμενη ηλικία συνταξιοδότηση που προβλέπεται από την Εθνική Νομοθεσία. Κάποιοι νομίζουν ότι η ηλικία συνταξιοδότησης ε, και η ηλικία του πότε βγαίνει κανείς σε σύνταξη, δηλαδή πότε παίρνει τη σύνταξη και πότε βγαίνει στη σύνταξη, δεν ταυτίζονται οι δύο αυτές ε, ηλικίε, αν θέλετε. Δηλαδή, νομίζω ότι ο καθένα μπορεί να βγει στη σύνταξη όποτε θέλει. Και όποιο θέλει να δουλέψει πιο πολύ, να μπορεί να δουλέψει πιο, για πιο πολλά χρόνια. Η συμβαστική Q δεν καλύπτει βέβαια όλη την τροπολογία μου 233, αλλά νομίζω ότι ε, στο και ως ένα βαθμό αποτελεί να βήμα προς την σωστή κατεύθυνση, όπως είπε και ο κύριος Ντίοντεν, γιατί μιλάει για το ξεκίνημα μια συζήτησης, ενός διαλόγου, άρα μπορώ τελικά να υποστηρίξω τη συμβιβαστική Q. Κάποια στοιχεία όμως τα οποία θα πρέπει να έχετε υπόψη, οι περισσότεροι γνωρίζετε για τις τροπολογίες ΕΚΟΝ ότι είναι αποδεκτές χωρίς ε, ψηφοφορία υπό ε, το άρθρο 50, άρα ψηφίζουμε. Δεν ψηφίζουμε στις τροπολογίες αυτές, παρότι πολλοί τι σχολίασαν. Επίσης, μέχρι τις 11.30 μπορείτε να αντιδράσετε ε, σε σχέση με τον τελικό κατάλογο ψηφοφορίας, τον οποίο έχετε λάβει σήμερα το πρωί. Και τώρα, πάρα πολύ γρήγορα, θα δώσω το λόγο στην Όμεν Ρόιτεν, γιατί έχουμε και την έκθεση Κοφεράτη. Πόσο χρόνο έχω στη θέση μου, λέει η κυρία Όμεν, 10 λεπτά. Καταρχήν, να σας ευχαριστήσω. Εγώ αυτό που ήθελα είναι περισσότερη ευελιξία όσον αφορά την ηλικία συνταξιοδότηση. Οι νέοι συνάδελφοι στην Βουλή της Ολλανδίας ζητάνε ευελιξία για το θέμα αυτό. Στην Ευρώπη είμαι σίγουρη ότι η συζήτηση αυτή δεν θα σταματήσει. Θα συνεχίσω στα Ολλανδικά κυρία Γκέρλινγκ. Μας λέτε ότι δεν επιθυμείτε να καθοριστούν δείκτες στην Ευρώπη όσον αφορά την αποδεκτή σύνταξη, το αποδεκτό επίπεδο σύνταξη. Εγώ διαφωνώ σε αυτό. Καθότι θεωρώ ότι οι κοινωνικοί εταίροι και τα κράτη-μέλη αλλά και οι ενώσεις των ε, συνταξιούχων θα πρέπει από κοινού να οργανώσουν ε, μία διαβούλευση και να καθοριστούν αυτά τα επίπεδα. Βεβαίως αυτό μπορεί να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα του κάθε κράτους μέλους και ο πρώτος πυλώνας θα πρέπει έτσι κι αλλιώς να κάνει μία αποδεκτή πρόταση. Δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να επιβάλλει ένα επίπεδο ευρωπαϊκό. Μιλάμε λοιπόν για αποδεκτό επίπεδο βάσει του πρώτου πυλώνα. Και βεβαίως μπορεί αυτή η συμβαστική λύση να γίνει ακόμα πιο αποδεκτή. Κυρία Φιγκερέιντο, και εγώ έχω κάποιες επιθυμίες και προτάσεις. Όμως, όμως, ξέρετε πολύ καλά ότι η πυραμίδα, η ηλικιακή πυραμίδα έχει αλλάξει στην Ευρώπη. Εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι είναι πολύ σημαντικός ο πρώτος πυλώνας. Σήμερα έχουμε όμως πολύ λιγότερους νέους που συνεισφέρουν και χρηματοδοτούν το σύστημα. Έχει αυξηθεί ο αριθμός των ηλικιωμένων, οι οποίοι ζουν πολύ περισσότερο. Οι νέοι σήμερα φτάνουν στην αγορά εργασίας πολύ αργότερα. Αυτό αποδυναμώνει τον πρώτο πυλώνα. Έχει αντιστραφεί η ηλικιακή πυραμίδα και εσείς δεν κάνετε απολύτως καμία ε, πρόταση. Αυτό μου φαίνεται παράδοξο. Γιατί από τη μία διαπιστώνετε αυτή την αλλαγή, από την άλλη δεν κάνετε καμία πρόταση. Αυτό δεν είναι σωστό. Κυρία Φικερέντο, το μέλλον των συνταξιούχων θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και ακόμα και αν δεν συμφωνώ με τις προτάσεις πρέπει να συνεργαστούμε Κυρία Κονέλισεν, πού δεν υπάρχει επικουρικότητα, ιδιαίτερα για θέματα προσδόκιμου ζωής, παραδείγματος χάρη, ηλικίας. Η επικουρικότητα είναι καθοριστική στον τομέα αυτό. Όπως είπα λοιπόν, για την ηλικία συνταξιοδότησης πρέπει να υπάρξει διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και αυτό να καθοριστεί ανακράτος μέλος. Τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία θα πρέπει να αποφασίσουν αν ναι ή όχι θα αυξήσουν το επίπεδο. Βεβαίως, ο καθένας μπορεί να αποφασίσει ότι, παραδείγματος χάρη στη Βουλγαρία, το όριο της συνταξιοδότησης είναι 65 στο 65ο όριο ε, έτος της ηλικίας, συγγνώμη. Εάν όμως το προσδόκιμο ζωής είναι 68, καταλαβαίνετε ότι εδώ μπορεί να υπάρχει ένα πρόβλημα. Μου λέτε όμως ότι δεν υπάρχουν κοινωνικές εγγύησεις Ζητώ συγγνώμη, αλλά εάν υπάρχει κάποιος που θεωρεί πολύ σημαντικό το θέμα των κοινωνικών εγγύσεων, είμαι εγώ σε αυτή την Επιτροπή. Δεν δέχομαι λοιπόν αυτή την παρατήρηση. Σας ευχαριστώ κύριε Πράνταν για τις παρατηρήσεις σας. Το θέμα της ηλικίας είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα. Γι' αυτό και προσπάθησα να το εξετάσω πάρα πολύ προσεκτικά, έτσι ώστε και το ΕΛΚ και οι φιλελεύθεροι να στηρίξουν αυτή την συμβιβαστική πρόταση. Λέτε ότι θα το στηρίξετε. Χρειάζεται όμως μια βάση πάνω στην οποία να συζητήσουμε. Προσπαθώ να πλησιάσω τη δική σας θέση, βεβαίως διατηρώντας ολόκληρο τον ιστό των προτάσεών μας. Όσον αφορά την τροπολογία της κυρίας Λίν και αυτή την πήρε υπόψη μου. Για τον πρώτο πυλώνα, όντως έκανα πολύ λίγες παρατηρήσεις για να μπορέσω να στηρίξω το αρχικό κείμενο. Κυρία Πρόεδρε, η παράγραφος 5 που επίσης ανέφερε και ο κύριος Ερή. Πρέπει να ανταμείψουμε τα κράτη-μέλη τα οποία δραστηριοποιούνται έτσι ώστε να δημιουργήσουν ένα βιώσιμο σύστημα. Αυτό είναι θετικό και νομίζω ότι σε αυτό συμφωνούν όλοι. Όμως, εσείς μας λέτε ότι το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης δεν μπορεί να αλλάξει και ότι η Επιτροπή, η Οικονομική Επιτροπή θεωρεί ότι πρέπει να ξανασυζητήσουμε αυτά τα σημεία. Εγώ στα σημεία 9 και 10 θεωρώ ότι επαναλαμβάνουμε τα ίδια. Γι' αυτό και στην παράγραφο 5, και αυτό δεν είναι μόνο δική μου άποψη, θεωρώ ότι αρκεί. Βεβαίως, εάν επιμένει η Οικονομική Επιτροπή, μπορούμε να επανέλθουμε, γιατί επαναλαμβάνω τα σημεία 2, 9 και 10 δεν ε, μπορούν εδώ να συμπεριληφθούν χωρίς να πλήξουμε τη συνοχή του κειμένου. Στον κύριο Έρη θα πω ότι πολλές χώρες δεν έχουν λάβει καθόλου υπόψη τους ποτέ τον πυλώνα 2. Γιατί, διότι τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είχαν κάποιες προτάσεις για τις συντάξεις. Τι έκαναν τότε τα κράτη-μέλη. Πήραν ένα τμήμα της δημόσιας χρηματοδότησης και κάποια, κάποιους άλλους πόρους από τον ιδιωτικό τομέα και δημιούργησαν ένα δεύτερο πυλώνα, ο οποίος δεν ήταν δεύτερος πυλώνας, ήταν ένας πυλώνας ε, ένα αλφα θα έλεγα. Η Ουγγαρία τι έκανε. Πήρε τα χρήματα αυτού του πυλώνα 1α και τα μετέφερε στον πυλώνα 1. Επί ένα χρόνο, επί ένα χρόνο, εποφελείται η Ουγγαρία. Αυτό κάνει. Από αυτή τη χρηματοδότηση. Και δεν υπάρχει απολύτως καμία πληρωμή. Καθυστέρηση λοιπόν ενός χρόνου. Στην Μαρία Νάρκιν θα ήθελα να πω ότι την ευχαριστώ πάρα πολύ για τα θετικά της σχόλια. Εγώ προσπάθησα να βρω μια σωστή διατύπωση. Αν έχετε κάποια πρόταση μπορείτε να μου την υποβάλλετε. Σας ευχαριστώ. Η παράγραφος 9 της Οικονομικής Επιτροπής συμφωνώ μαζί σας ότι θα πρέπει να αναδιατυπωθεί. Αλλά ελάτε να προσπαθήσουμε να βρούμε μαζί μια καλύτερη διατύπωση. Γιατί εγώ τελικά τι ήθελα να εκφράσω στην παράγραφο αυτή. Θέλησα, παραδείγματο χάρη, να δημιουργήσω ένα μεγάλο οριζόντιο συνταξιοδοτικό ταμείο. Ένα μεγάλο συνταξιοδοτικό ταμείο, το οποίο σε περιφερειακό επίπεδο ή τοπικά να μπορούν να συνεισφέρουν. Αυτό ήθελα να πω. Τώρα, αν η διατύπωση δεν είναι σαφής, πραγματικά μπορούμε να το ξαναδούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνεργασία σας και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όσον αφορά τη συνοχή του κειμένου, ιδιαίτερη της τροπολογίας κυρίας Έκον. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρε. Περνάμε στο... Στην έκθεση του κύριου Κοφεράτη, σε σχέση με συνέργειες μεταξύ του Περιφερειακού Ταμείου και του Κοινωνικού Ταμείου, σας ευχαριστώ πρόεδρε λέει ο Κομφεράτη. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα Κοίτα. να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους οι οποίοι κατέθεσαν τροπολογίες γιατί έδειξαν μεγάλη διαθεσιμότητα να αναζητήσουν αποτελεσματικές συμβαστικές λύσεις μαζί μου και νομίζω ότι το έργο το οποίο κάναμε από κοινού ήταν ένα εποφελές έργο με το οποίο μπορούμε να καταλήξουμε σε μια συνενετική απόλυξη. Γνωρίζετε το στόχο αυτού του εγχειρήματο γιατί έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν. Θέλουμε να τονίσουμε την αποτελεσματικότητα των διαρθρωτικών ταμείων, να προσπαθήσουμε να δώσουμε μεγαλύτερη ορατότητα στη δράση του με ε, συγκεκριμένους κανονισμούς και πόρους που πηγαίνουν σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις και ιδίω να τονώσουμε τον προβληματισμό που μπορεί να οδηγήσει σε μια μεταρρύθμιση των ταμείων αυτών στο μέλλον. Νομίζω ότι αυτό το πλαίσιο ήταν κάτι το οποίο έγινε δεκτό σε γενικές γραμμές από όλους και οι θέσεις των διαφόρων συναδέλφων το καταδεικνύουν. Το πιο αμφιλεγόμενο τώρα σημείο, χωρίς να ανατρέπει το γενικό πλαίσιο της σκέψης μας, είναι το θέμα του μέλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Γιατί υπάρχει και το σενάριο στην ε, συμβαστική τροπολογία που παρουσιάστηκε να ζητήσουμε από την Κομισιόν να υπάρξει μια αύξηση της χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για τα επερχόμενα έτη ενώ παράλληλα αυτή η δυνατότητα αύξησης χρηματοδότησης θεωρείται μη εφικτή από πολλούς άλλους και εξάλλου σε αντίφαση με την χρηματοδότηση των άλλων ταμείων. Εγώ νομίζω ότι είναι το μόνο σημείο το οποίο παραμένει επίμαχο μετά από τις συζητήσεις που κάναμε. Αν θέλουμε λοιπόν να ζητήσουμε την αύξηση της χρηματοδότησης μέχρι το 2020 που να έχει από τους θεμελιώδεις πυλώνες της την αύξηση της ε, απασχόλησης και ιδίω της ποιότητας της απασχόλησης και όχι μόνο του όγκου της απασχόλησης, δεν θα ήταν λαθασμένο να ζητήσουμε μεγαλύτερη χρηματοδότηση του κοινωνικού ταμείου που είναι ακριβώς αυτό το οποίο έχει την λειτουργία να προωθεί την απασχόληση. Τούτου λεχθέντος βέβαια, θα είναι τα συμπεράσματα τα οποία θα αντλήσουμε και θα αντλήσουν οι λήπτες αποφάσεων για τη χρηματοδότηση αυτή, αλλά εναπόκειται πιστεύω και στην Κομισιόν να καταλήξει σε μια δική της θέση και να παρουσιάσει τα συμπεράσματά της με ένα κείμενο το οποίο θα συμπεριλαμβάνει και τις απόψεις της δικής μας Επιτροπής, η οποία και δεν είναι τυχαία, έχει μεγάλη ευαισθησία για τα θέματα απασχόλησης και εργασίας διότι τα έχουμε αντιμετωπίσει σε όλες τις διάφορες και πολυπίκυλες πτυχές τους. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω τους συναδελφούς για τη συμβολή που έκαναν στην εκπόνηση αυτής της νομοδότησης. Νομίζω ότι το έργο στο οποίο απεδίθησαν ήταν αποτελεσματικό και εξάλλου το θέμα αυτό θα είναι σημαντικό να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε με μια σύγκληση απόψεων, κάτι το οποίο δεν αποκλείεται, αλλά θα ήταν πάρα πολύ θετικό να υπάρξουν κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ, λέει και η Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την συνεργασία. Νομίζω ότι πραγματικά είναι πολύ καλή η συμβαστική λύση. Μπορέσαμε να συμπεριλάβουμε πολλές τροπολογίες και βρισκόμαστε, θα έλεγα, στην σωστή κατεύθυνση. Εν πάση περιπτώσει, μπορούμε εδώ να προτείνουμε μια καλή λύση επικοδομητική και να λάβουμε υπόψη μας ε, και τα διάφορα συνταξιοδοτικά συστήματα, να λάβουμε υπόψη μας τις διαφορές, κάποια ευελιξία και βεβαίως να δούμε ποιοι είναι οι οργανισμοί αυτοί χρηματοδότησης ε, επιτόπου να υπάρξει η χρηματοδότηση χωρίς να υπάρχουν δυσκολίες όσον αφορά την ροή των πόρων. Νομίζω λοιπόν πραγματικά ότι κάναμε ένα καλό βήμα, θετικό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 Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή, ιδιαίτερα για τις συμβιβαστικέ του τροπολογίες, οι οποίες πραγματικά είναι πολύ και συμφωνώ με την προηγούμενη ομιλήτρια. Είναι πολύ χρήσιμη και ουσιαστική η έκθεση αυτή και είμαι πεπισμένος ότι πρόκειται για ένα πακέτο συμβαστικό το οποίο πραγματικά θα μπορέσουμε να στηρίξουμε. Συμπεριλαμβάνει πάρα πολύ καλές λύσεις και προτάσεις και θα ήθελα να συμπεριλάβω κάτι. το οποίο θα μπορούσαμε να σκεφτούμε σήμερα κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης. Πρόκειται για τη συμβιβαστική τροπολογία F σε αυτήν την συμβαστική τροπολογία αναφέρεται το θέμα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, των πόρων που θα πρέπει να αυξηθούν. Κατά την άποψή μου υπάρχουν εδώ δύο δυσκολίες. Από τη μία, κάτι το τυπικό. Όχι τόσο πολύ επί της ουσίας, Τη συμβαστική τροπολογία υπάρχει πρόβλημα. Μιλάμε για τη στρατηγική για το 2020 και αν θέλουμε να λάβουμε υπόψη μα και όλε τι συνέπειε αυτή τη οικονομική κρίση, θα πρέπει να δούμε πώ μπορούμε να δημιουργήσουμε θέσει απασχόληση. Πώ μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα και να ξεπεράσουμε την κρίση εάν δεν μειωθεί η ανεργία και δεν δημιουργήσουμε νέες θέσεις απασχόλησης. Αυτός ο στόχος δεν μπορεί να επιτευχθεί αποκλειστικά και μόνο μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Δεν είναι το μόνο εργαλείο που διαθέτουμε. Θεωρώ λοιπόν ότι θα ήταν πολύ πιο επικοδομητικό να πούμε όλα τα ταμεία συνοχής των οποίων οι πόροι θα πρέπει να αυξηθούν για να δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης. Δεύτερον, μέτρα επαγγελματικής κατάρτισης, τα οποία θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν από τα ευρωπαϊκά ταμεία και θα πρέπει να βρούμε τρόπους να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων, να στοχεύσουμε σωστά οι ανησυχίες αυτές θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Νομίζω θα πρέπει οι πολιτικές ομάδες να σκεφτούν όλα αυτά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να συμβαστώ αυτά που είπε ο κύριος Κομφεράτη, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και είναι σημαντικό να έχουμε και τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εν ώψη της νέας περίοδου προγραμματισμού θέλω να υπογραμμίσω δύο σημεία σε σχέση με τον προβληματικό χαρακτήρα που έχει η κοινωνική κατάσταση σε πολλές χώρες μεταξύ των οποίων και της δικής μου. Δύο προβλήματα. Πρώτον, η τωρινή κρίση και οι δυσκολίες που υπάρχουν σε πολλά κράτη-μέλη έχει σαν αποτέλεσμα σε πολλές χώρες πολλά προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, παραδείγματος περιφερειακά ή επαρχιακού επίπεδου, δεν έχουν υλοποιηθεί. Δεν υπήρχαν ακόμα και αιτήσει για να προγραμματιστούν τέτοιου είδου ενέργειε στα κράτη-μέλη, γιατί είτε τα κράτη-μέλη είτε οι περιφέρειες σε ορισμένε χώρε που έχουν αποκεντρωμένο σύστημα δεν έχουν επαρκεί πόρου συγχρηματοδότηση αυτών των προγραμμάτων για τα κοινωνικά θέματα σε εθνικό, σε περιφερειακό επίπεδο και έτσι τα προγράμματα αυτά δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Το τονίζω σε αυτή την κατάσταση είναι πάρα πολλέ χώρε. Ίσως και εδώ η Κομισιόν θα μπορούσε να αναλάβει κάποια πρωτοβουλία να μας παρουσιάσει την κατάσταση αυτή θα ήταν χρήσιμο. Μάλλον η δική μας Επιτροπή να οργανώσει μια ακρόαση μαζί με την Επιτροπή Περιφερειακών Υποθέσεων για να καταλάβουμε καλύτερα σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Πριν από το τέλος της περίοδου προγραμματισμού που τελειώνει το 2013 σε σχέση με την εκταμείευση των ταμείων των ποσών από τα ταμεία αυτά. Δεύτερον, σε πολλές χώρες επιτρέπεται κάτι, το να χρησιμοποιηθεί δηλαδή το κοινωνικό ταμείο για να γίνουν ενέργειες οι οποίες αντιμετωπίσουν επίγοντα πρόβλημα απασχόλησης, δηλαδή για να δημιουργηθούν κατά κάποιο τρόπο κοινωνικά δίκτυα ασφάλειας στα κράτη-μέλη, να βοηθηθούν άτομα τα οποία ε, είναι άνεργοι κτλ. Αυτό όμως έχει προβλήματα, ενώ είναι κατανοητή αυτή η ενέργεια, αυτό ουσιαστικά περνάει τη χρήση του κοινωνικού ταμείου από την χρήση του για την κατάρτιση και τη δημιουργία νέων δεξιοτήτων, ουσιαστικά το περνάει σε μια άλλη φάση που είναι απλώς αντιμετώπιση της ε, χρηματοοικονομικής κρίσης. Το ξέρω γιατί αυτά τα νέα στοιχεία έχουν δημιουργήσει προβλήματα στη διαχείριση των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είναι λοιπόν ζητήματα τα οποία θα πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας και το θέμα αυτό πρέπει να συνεχίσει να απασχολεί την Επιτροπή μας, αλλά ίσως πρέπει να συνεργαστούμε σε μια κρόση με την Επιτροπή των Περιφερειακών Υποθέσεων. Ευχαριστώ. Πίσω στον κύριο Κοφεράτη για να συνοψίσει. Ταχύτατος και τηλεγραφικός θα είμαι. Είναι φανερό ότι ο χρόνος που μας ε, χωρίζει από την απογευματινή ψηφοφορία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αυξήσουμε ακόμα περισσότερο το βαθμό συνένεσης σε σχέση με το πλαίσιο το οποίο έχω παρουσιάσει, συμβαστικές τροπολογίες κτλ. Σε ό,τι αφορά στην διάσταση της χρηματοδότησης, εγώ δεν πιστεύω στο σενάριο αυτό βάσει του οποίου η αύξηση των κονδυλίων του Κοινωνικού Ταμείου θα πρέπει να είναι σε βάρος των άλλων διαρθωτικών ταμείων. Αυτό θα ήταν ένα πολύ σοβαρό λάθος. Εγώ πιστεύω ότι είναι απαραίτητο τα διαφθορτικά ταμεία στο σύνολό τους να τύχουν αύξηση κονδυλίων και μέσα σε αυτή την αύξηση να δοθεί ιδιαίτερη μέρημνα στην αύξηση των πόρων του Κοινωνικού Ταμείου, γιατί είναι αυτό το οποίο εμπλέκεται ιδιαίτερα με τα θέματα απασχόλησης. Κατανοώ τώρα τις ανησυχίες των συναδέλφων από το ΕΛΚ, αλλά θέλω να τους καθησυχάσω. Αν χρειάζεται μια διευκρίνηση μπορούμε να το κάνουμε και στο κείμενο. Αλλά κανείς από μας δεν θεώρησε ότι η ενίσχυση του κοινωνικού ταμείου θα πρέπει να γίνει σε βάρος των άλλων ταμείων. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Επίσης ξέρω πώς χρησιμοποιούνται οι πόροι του κοινωνικού ταμείου σε πολλές χώρες όπως η δική μου. Όχι μόνο αυτά που είπε η κυρία Κώστα ότι υπάρχει δυσκολία της συγχρηματοδότησης, αλλά επίσης και η έλλειψη χρησιμοποίησης του Κοινωνικού Ταμείου και που πολλές φορές χρησιμοποιείται σαν υποκατάστατο των κοινωνικών δικτύων ασφαλείας που δεν λειτουργούν σε πολλές χώρες. Το ουσιαστικό σημείο είναι το θέμα της κατάρτισης. Είναι προφανές ότι όταν χάνει κανείς τη θέση εργασίας του είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσει να μπει σε ένα σύστημα κατάρτισης και για αυτή την κατάρτιση προφανώς μπορεί να παρέμβει το κοινωνικό ταμείο. Αυτό όμως το οποίο δεν θεωρώ ότι είναι αποδεκτό είναι ορισμένες φορές η κατάρτιση αυτή να είναι πλασματική. Δηλαδή να έχει χαρακτήρα μαϊμούς και να μην έχει σαν στόχο την ανύψωση των επαγγελματικών κριτηρίων των ε, ανέργων, αλλά απλώς να είναι ένα πρόσχημα για να δοθεί κάποιο εισόδημα στα άτομα αυτά. Με κάθε κατανόηση για την κατάσταση των ανθρώπων οι οποίοι έχουν χάσει τη θέση εργασίας τους και τις δυσκολίες και του ευαίσθητου χαρακτήρα του, ε, της κοινωνικής του κατάστασης, τέτοιου είδους δράσεις θα πρέπει να αποθαρρυνθούν και να είναι σαφές αυτό και από τους κανονισμούς του κοινωνικού ταμείου. Αυτό είναι ένα εκφυλιστικό φαινόμενο το οποίο δεν πρέπει να το αποδεχτούμε και όταν υπάρξει αναθεώρηση του κανονισμού θα πρέπει να έχουμε ε, στο μυαλό μας ότι πίσω από την ίδια λέξη κατάρτιση μπορούν να υποκρύπτονται πάρα πολλά πράγματα. Thank you very much. And the vote, you know, Ευχαριστώ. Σήμερα το απόγευμα ψηφίσουμε όπως ξέρετε. Ευχαριστούμε κύριε Κοφράτη. Περνάμε Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Σύραξης. Ο κύριος Κάσλερ έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κηρύξει, θέλει να κηρύξει το έτος 2012 έτος ενεργούς γύρανσης με τρόπο ώστε να προσελκύσει την προσοχή της κοινή γνώμη στο θέμα αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό και να υπάρξει η σύνδεση της ενεργούς γύρανση με τις δυνατότητε καλύτερη απασχόλησης σε επίπεδο ποιότητα και τι δυνατότητε δράσης για, την, για τις πιο μεγάλε ηλικίε στην Ευρώπη. <clears throat> Το ευρωπαϊκό αυτό έτος θα πρέπει να υπογραμμίσει και να τη σημασία της συμβολής της τρίτης ηλικίας στον χώρο εργασίας και να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη και η γενιά 55 χρόνων και πάνω να ενισχυθεί. Η επιλογή αυτού του θέματος λοιπόν δεν είναι ξένη με πολλές συζητήσεις που είχαμε εδώ στην Επιτροπή Απασχόλησης. Μιλήσαμε για το γεγονός ότι πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία μεταξύ των γενεών. Εγώ θέτω το ερώτημα με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε πέραν αυτής της γκρίζας γενιάς ή ασημένιας γενιάς άμα θέλετε να δούμε και άλλες πτυχές της αγοράς εργασίας που συνδέονται με τους νέους. Δηλαδή να φτιάξουμε μια γέφυρα αλληλεγγύης μεταξύ των γενναίων. Αν το πιστεύουμε, και αυτό νομίζω ότι έχει δείξει και η συζήτηση στην Επιτροπή μας με ε, εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, όταν συζητάμε με το θέμα της ε, ενεργούς ε, γύρανσης, Το θέμα αυτό <clears throat> και από την πλευρά των εργοδοτών και των εργαζομένων θα πρέπει να συνδεθεί με το θέμα της αλληλεγγύης μεταξύ των γενναίων. Επομένως, η πολιτική αυτή διάσταση της ε, αγοράς αντιμετωπίζεται από την ε, Επιτροπή με έναν τρόπο που δεν είναι πανταφεντικό με την έννοια τη απασχολησιμότητας. Εμείς όμως θα πρέπει να προσθέσουμε μια κοινωνική διάσταση σε αυτή την προβληματική και κυρίω την αλληλεγγύη μεταξύ των γενναιών μέσα στο έτος 2012 που θα είναι το έτος ενεργούς γύρανσης και για μένα πρέπει να προσθέσουμε και την αναγνώριση των ε, προσφορών που έχουν κάνει τα άτομα τα οποία έχουν εργαστεί μέχρι μια μεγάλη ηλικία, τα οποία και στον τομέα των οικογενειακών και στον τομέα της εργασίας συνεχίζουν μέχρι μια μεγάλη ηλικία αλλά επίσης θα πρέπει να περιλάβω με μια τροπολογία, θα το υποβάλω αυτό και στην εκθεσή μου, να περιληθούν και αυτοί οι οποίοι φροντίζουν άτομα τα οποία είναι ανήμπορα ή ε, έχουν αναπηρίες. Ο στόχος μου λοιπόν θα είναι να έχουμε μια κοινή αντιμετώπιση, όχι μονάχα δηλαδή την ενεργογύρανση, αλλά και μια κουλτούρα ενεργούς ε, γύρανσης, να δώσουμε έμφαση στην ε, ζωτικότητα και στην υγεία σε μεγάλη ηλικία. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία συμβάλλουν στην αξιοπρέπεια του ανθρώπου και στην αλληλεγγύη μεταξύ των γενναιών. Και πρέπει να είναι στο προσκήνιο, επομένω. Κάτι το οποίο είναι επίση σαφέ και είναι ένα σημείο το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε σήμερα μεταξύ μα και το οποίο έχουν αντιμετωπίσει και άλλε επιτροπέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ότι χρειάζεται ένα δεσμευτικό προπολογισμό για το έτο αυτό το 2012 τη η, η δική μου έκθεση προτείνει 6 εκατομμύρια ευρώ. Η Περιφερειακή Επιτροπή έχει προτείνει 8 εκατομμύρια νομίζω. Μπορούμε να συζητήσουμε για τον προπολογισμό αυτό. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι να μπορέσουμε να έχουμε μια επικοδομητική αντιμετώπιση μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για να καθορίσουμε ένα συγκεκριμένο ποσό για τον προπολογισμό του έτου 2012. Ελπίζω λοιπόν ότι αυτό με υποστηρίζει σε αυτό η πλειοψηφία, αν όχι όλοι σα, ότι θα πρέπει το ταχύτερο δυνατό να αργωνώσουμε αυτό το έτος 2012 γιατί είναι ουσιαστικά σε 11 μήνες από σήμερα. Είναι απαραίτητο να το κάνουμε έτος ευαισθητοποίησης κοινή γνώμης για το θέμα της ενεργούς γύρανσης και επομένως σιγά σιγά θα πρέπει να κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες και να επιταχύνουμε τη δράση μας. Ένα τελευταίο σημείο το οποίο για μένα είναι επίσης πολύ σημαντικό είναι η τήρηση της αρχής της επικορικότητας η οποία πρέπει και αυτή να γίνει αναγνωριστή μέσα στην πρόταση της Κομισιόν και στη δική μου έκθεση τονίζεται ότι το έτος αυτό δεν είναι έτος για μια νέα νομοθετική δράση, αλλά είναι έτος ευαισθητοποίησης και επομένως θα είναι πιο εύκολο για όλους να συμφωνήσουν σε αυτή την κατεύθυνση, εφόσον δεν πρόκειται για νέα νομοθεσία. Περιμένω λοιπόν να ακούσω τις απόψεις των συναδέλφων και θέλω να ευχαριστήσω και την ε, Κομισιόν και το Συμβούλιο για τις άτυπες ε, συζητήσεις που είχαμε και τη συνεργασία τους όπως και της γραμματείας και τους ε, σκιώδεις εισηγητές θέλω να ευχαριστήσω και θέλω να τους παρακαλέσω όσο το δυνατόν πιο γρήγορα μετά από αυτή τη συζήτηση να προχωρήσουμε σε διαπραγματεύσεις ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε σάρκα και ωστά στο έτος 2012 για μια κουλτούρα ενεργούς γύρανσης και ζωτικότητας και δράσης. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Σάντα από την Ουγγρική Προεδρία. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας καλωσορίζω όλους. Η Προεδρία σας ευχαριστεί πολύ για την πρόσκληση να συμμετέχουμε κι εμείς στην σημερινή συζήτηση. Θέλω να σας πω ότι το Συμβούλιο έχει ήδη προετοιμάσει μία θέση για την έκθεση του κ. Κάρστεν και βεβαίως είδαμε με μεγάλη χαρά την πρόταση της Επιτροπής να γίνει το 2012 το Ευρωπαϊκό Έτος για την Ενεργογύρανση. Το Συμβούλιο ήδη από τις 6 Δεκεμβρίου του 2010 έχει εκφράσει την άποψή του για το θέμα αυτό και έχουμε θέσει σαν στόχο, σαν συμβούλιο, να συμφωνήσουμε ήδη από την διαδικασία της πρώτης ανάγνωσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εξ λοιπόν της Προεδρίας του Συμβουλίου θα ήθελα να σας πω ότι θα θέλαμε να συνεργαστούμε με τον εισηγητή για να επιτύχουμε τον στόχο μας. Ήδη έχει ξεκινήσει μια πρώτη συζήτηση για την έκθεση και θεωρούμε ότι είναι μια πολύ καλή βάση η υπάρχουσα έκθεση για την συνέχιση της ε, συζήτησής μας. Υπάρχουν δύο σημεία τα οποία ακόμα ε, χρειάζονται συζήτηση και επεξεργασία. Παρ' όλα αυτά θεωρούμε ότι η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να ε, επιτύχουν συμφωνία. Το... Τα ανοιχτά θέματα που θέλουν ακόμα συζήτηση είναι ο προπολογισμό και ο τίτλος. Το Συμβούλιο λοιπόν έχει δεσμευθεί να συμφωνήσει με το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή των Συντοματών Δυνατών έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να αναλάβουν τις πρωτοβουλίες προετοιμασίας για το έτος 2012, έτος της ενεργούς γύρανσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χιάκοπ, εξ ονόματος Επιτροπής, έχει το λόγο. Uh, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τον εισηγητή αλλά και στους υπόλοιπους βουλευτές οι οποίοι ε, μας ε, έδειξαν ότι στηρίζουν την πρότασή μας για ένα ευρωπαϊκό έτος ενεργού γύρανσης. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό από τη σκοπιά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να γίνει γρήγορα δεκτή η πρόταση αυτή ώστε να ε, στείλουμε ένα πολύ ηχηρό μήνυμα σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς για το ευρωπαϊκό αυτό έτος ώστε να ξεκινήσουν να προετοιμάζουν τις πρωτοβουλίες και για να στεφθεί έτσι και με επιτυχία αυτό το ευρωπαϊκό έτος. Αυτό που μας μας φοβίζει περισσότερο είναι πως υπάρξει κάποια εμπλοκή μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων που είναι αρμόδια για τον προπολογισμό σε ό,τι αφορά ακριβώς τον προπολογισμό. Δηλαδή Συμβούλιο και Κοινοβούλιο μπορεί εκεί να ε, συγκρουστούν ίσως, ε, να μην συμφωνήσουν. Θα πρέπει πάντως να είναι σαφής η δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Ευρωπαϊκό έτος και στο χρηματοοικονομικό επίπεδο. Και αν θα ήθελα να πω εν συντομία στην Επιτροπή σας ότι έχουμε πόρους στη διάθεσή μας συγκεκριμένα από τον προπολογισμό του 2011, που είναι ένας πολύ κρίσιμος προπολογισμό, γιατί τα χρήματα τα οποία έχουν δεσμευτεί το 2011 θα δώσουν αποτελέσματα, πραγματικά αποτελέσματα στη διάρκεια του ευρωπαϊκού έτους. Τώρα, και επιπλέον πόροι από τον προπολογισμό 2011, ίσως, 2012, ίσως να μην κάνουν και μια σημαντική διαφορά λόγω του χρόνου που θα χρειαστεί για να φτάσουν οι πόροι αυτοί στους δικαιώχους και να χρησιμοποιηθούν για συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Τώρα, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη και την επιθυμία του Κοινοβουλίου να φανεί ότι υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι για το ευρωπαϊκό έτος, ίσως ε, μία λύση θα μπορούσε να είναι όχι να έχουμε ένα άρθρο το οποίο θα απαιτεί μια νέα συγκεκριμένη θέση του προπολογισμού για το ευρωπαϊκό έτος, αλλά μια αιτιολογική σκέψη η οποία θα αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη δεσμεύει κάποια χρήματα για το ευρωπαϊκό έτος. Είμαστε λίγο στα 4, γύρω στα 4 εκατομμύρια. Αυτό είναι το διαθέσιμο ποσό, λίγο πάνω, λίγο κάτω, για ένα κονδύλιο του προπολογισμού. Ζητήσαμε να αυξηθεί ε, η προκοδότησή του για το 2011 και θα ζητήσουμε το ίδιο και για το 2012, ώστε να υπάρχει αυτό το ποσό διαθέσιμο. Και το ποσό αυτό δεν απέχει και τόσο από την αρχική πρόταση του εισηγητού. Βέβαια, σίγουρα υπολείπεται σε κάποιο βαθμό του ποσού που ζητεί η Περιφερειακή Επιτροπή. Φυσικά μπορούμε να διατυπώσουμε μία πρόταση σύνταξης και έτσι θα μπορέσουμε να αποφύγουμε να υπάρξει και αυτή η αντιπαράθεση Κοινοβουλίου με Συμβούλιο. Πρώτα, σας ευχαριστώ πολύ. Πρώτος ομιλητής, ο κύριος Κάση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ την Ουγγρική Προεδρία, ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχάς θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή, αλλά να πω συγχρόνως ότι υπάρχουν και κάποια θέματα που εκ μέρους της Άλντε θα ήθελα να σας αναφέρω. Η αρχική πρόταση βασιζόταν σε πολύ μεγάλο βαθμό στην επιμήκυνση ε, της οικονομικής δραστηριότητας ε, για μεγαλύτερη ηλικία. Η ενεργο γύρανση ουσιαστικά νομίζουμε ότι πιο πολύ σημαίνει να παραμείνει κάποιος οικονομικά δραστήριος. Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι η οικογενειακή διάσταση, η δεύτερη δηλαδή διάσταση προστέθηκε, ο ρόλος που έχουν οι ηλικιωμένοι για την ανατροφή παραδείγματος χάρη των ε, παιδιών. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να αναφερθεί και θα ε, μας ικανοποιήσει ιδιαίτερη προσθήκη της οικογενειακής ε, ζωής. Αλλά πρέπει να μπει και μια τρίτη διάσταση, κοινωνικές δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν ούτε στο πλαίσιο της οικογενειακής ζωής, ούτε όμως φέρουν κάποιο εισόδημα. Όλα αυτά είναι σημαντικός παράγοντας για την υγιή και ενεργό γύρανση που θέλουμε να προωθήσουμε και να στηρίξουμε για τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας. Η συμμετοχή στον πολιτιστικό βίο, αθλητισμός, η εκπαίδευση πανεπιστήμια της τρίτης όπω όπως τα λέμε. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά στοιχεία για τι ζωέ των ηλικιωμένων συμπολιτών που θα μπορούν έτσι να έχουν μία έμεση ή άμεση συμμετοχή στην κοινωνική ζωή. Μπορούν οι ηλικιωμένοι να βοηθήσουν με τι δεξιότητε με τι γνώσει του, να βοηθήσουν και του άλλου, αλλά και του εαυτού του, παραμένοντα υγιεί, ανεξάρτητοι και κοινωνικά ενεργοί και δραστήριοι για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ένα από τα μεγαλύτερα μηνύματα που μπορεί να στείλει η ενεργός γέννας είναι ακριβώς ότι ε, θεωρείται πολλές φορές και άδικα, χαρακτηρίζεται ως βάρος ε, ε, ο ηλικιωμένος για την κοινωνία και πρέπει να παραμείνει παρόλα αυτά σε καλή υγεία, σε οικονομική ευμάρεια και βέβαια πολλές φορές μιλάμε και για διαγενειακή αλληλεγγύη. Δεν πρέπει να ξεχνούμε όμως ότι η ηλικιακή ομάδα που θεωρούμε ηλικιωμένους ή γυράσκοντες έχουμε λίγο πολύ υγιείς και ενεργούς πολίτες, λιγότερο ή περισσότερο. Επομένως, είναι σημαντική και η αλληλεγγύη μεταξύ των γενών. για να παραμείνουν ενεργοί οι ηλικιωμένοι θα πρέπει όλοι να φροντίσουμε αυτοί που είναι λιγότερο ευνοημένοι να έχουν σταθερούς δεσμούς και να μπορούν να έχουν ε, τουλάχιστον τα προστοζήν. Μιλάμε για την κοινωνική ένταξη και σίγουρα τους ε, ενεργούς πολίτες τους εντάσσει πιο εύκολα η κοινωνία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον τίτλο του Ευρωπαϊκού Έτους 2012, αυτό θα το συζητήσουμε αφού καταθέσουμε τροπολογίες. Η Άλντε όμως δεν θα υποστηρίξει την πρόταση του εισηγητή, γιατί είναι πολύ μακροής ο τίτλος αυτός για τον ενεργό, αν πούμε ευρωπαϊκότητα για την ενεργό γύρανση και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενναιών, νομίζω αρκεί ως τίτλος. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής. Σάπρενοκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή τον Μάρτιν Κάσλα Νομίζω ότι είναι πολύ καλή η εργασία του και είναι μια πολύ θετική βάση για τις μελλοντικέ μας συζητήσεις. Και καταρχήν υποστηρίζω την έκθεση αυτή. Να υπογραμμίσω ορισμένε πτυχές τώρα. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε το ότι η γύρανση δεν αφορά μόνο τους ηλικιωμένους. Αλλά και όλη την κοινωνία και για μας ίσως και την πιο νέα ε, γενιά θα είναι ίσως πιο δύσκολη γύρανση από αυτούς που ήδη έχουν προχωρήσει στην ηλικία του. Πρέπει να υποστηρίξουμε επίσης και τη συμπερίληψη της ε, γενναίας των ηλικιωμένων στην αγορά εργασίας. Δεν πρέπει να τους υποχρεώσουμε να δουλεύουν. Αλλά θα πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να γίνει εφικτή η απασχόλησή τους και να μπορούν να πέσουν σημαντικό ρόλο στην αγορά εργασίας. Δεν θέλω να υπεραπλοποιήσω τα πράγματα. Νομίζω ότι αυτό όμως το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε την απαραίτητη ευελιξία στην αγορά εργασίας, να υπάρχουν ε, δυνατότητες εργασίας περιορισμένου χρόνου ή μονάχα σε σύντομα χρονικά διαστήματα, ώστε να συμπεριληφθούν περισσότερο και οι ηλικιωμένοι. Υπάρχει ο κίνδυνος να αποκλείονται λόγω του χάσματος πληροφόρησης. Πρέπει να βοηθήσουμε να, πάρουν, να έχουν περισσότερη πρόσβαση στις τεχνολογίες η πληροφόρηση και επικοινωνία, ώστε να μην έχουν να αντιμετωπίσουν το χάσμα αυτό πληροφορία, το οποίο του αποκλείει από την ενεργή ζωή στην κοινωνία μας. Υποστηρίζω επίσης και τα σχόλια σε σχέση με την σύνδεση μεταξύ του έτους ενεργούς γύρανσης με άλλα μέτρα και άλλα προγράμματα που πρέπει να είναι συνεχής και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη Ίσως η πτυχή της γύρανσης που έχει μεγάλη επίπτωση στη ζωή μας θα πρέπει να συνοδεύεται από διάλογο μεταξύ των γενεών και θα πρέπει να τονίσουμε την ανάγκη να έχουν πρόσβαση οι ηλικιωμένοι στις τεχνολογίες που τους βοηθούν να παραμείνουν ενσωματωμένοι στην κοινωνία και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ενεργό γύρανση. Επίσης πρέπει να αναγνωρίσουμε το ότι δεν μπορούμε να είμαστε αυτάρκεις και ε, ανεξάρτητοι μέχρι τον τάφο. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη ολοκλήρωση των κοινωνικών υπηρεσιών. Ευχαριστώ πολύ. Ο η Σίλβια Κώστα θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή γιατί είπε πολλά πράγματα Νομίζω ότι αυτό το οποίο είναι το ουσιαστικό το οποίο τονίστηκε ήταν η αλληλεγγύη μεταξύ των γενναίων που δείχνει και την πραγματική στοχοθεσία αυτού του έτους, του 2012 είναι προφανώς σημαντική λοιπόν η διατήρηση της ενεργητικότητας και της ζωτικότητας των ηλικιωμένων, όπως αναφέρεται στον τίτλο αυτού του έργου, του έτους μάλλον, αλλά θα πρέπει να κρατήσουμε στο προσκήνιο και τη σχέση μεταξύ των ε, γενναιών. Όχι μονάχα λοιπόν να είναι αποδέκτες παρεμβάσεων οι πιο ηλικιωμένοι, αλλά και ως ενεργός εμπλεκόμενοι στην αλληλεγγύη μεταξύ των γενναίων. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η αλληλεγγύη μεταξύ των γενναιών είναι μια προϋπόθεση για να υπάρξει ενεργός γύρανσης και πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να έχουμε αυτή την ολιστική προσέγγιση να αντιμετωπίσουμε και τα θέματα υγείας, την δυνατότητα να συνεχίσει η δραστηριότητα των ηλικιωμένων, τα θέματα πρόληψης για να μην υπάρξει μια γύρανση η οποία θα συνοδεύεται από ασθένειες. Πρέπει να συνδεθεί επίσης και με τη μείωση της και υπάρχουν και δύο ακόμα θέματα τα οποία πρέπει να συνδέσουμε. Το θέμα του εθελοντισμού, γιατί εφέτος είναι το έτος του εθελοντισμού. Να συνδέσουμε λοιπόν την διαδικασία του εθελοντισμού με τα ηλικιωμένα άτομα τα οποία με τις γνώσεις τους και την πείρα τους και τη σοφία τους μπορούν να προσφέρουν πάρα πολλά στην <clears throat> αν θέλετε επαγγελματικού χαρακτήρα εθελοντική δραστηριότητα και φυσικά μπορούν να παίξουν ένα παιδαγωγικό ρόλο, να βοηθήσουν σε κοινωνικό επίπεδο κτλ. Και ένα δεύτερο ζήτημα το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι να δείξουμε παραδείγματα προγραμμάτων και σχεδίων που ενθαρρύνουν αυτή την αλληλεγγύη μεταξύ των γενναίων... και καταδεικνύουν την πραγματικότητα των σχέσεων μεταξύ των γενναιών που πρέπει ήδη να τονίζεται και τα σχολεία και σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα σε πολλές ε, χώρες νέων που έχουν τα απαραίτητα προσόντα και οι οποίοι έχουν διδάξει τους πιο ηλικιωμένους πώς να χρησιμοποιούν τους κομπιούτερ. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να έχουμε και τη δυνατότητα της καινοτομία και της, πληροφο... της πληροφόρησης των ηλικιωμένων που μπορεί να έχει μεγάλη σημασία. Και ένα τελευταίο ερώτημα, πιστεύω ότι είναι σημαντικό να δώσουμε και μια ιδιαίτερη προσοχή μέσα στα πλαίσια της γνωμοδότησης Επιτροπής μας στην υποστήριξη πρέπει να δοθεί στις ΜΚΟ, στους φορείς, οι οποίοι προωθούν ακριβώς μια τέτοια προσέγγιση. Δηλαδή μια προσέγγιση η οποία δεν απομονώνει τους ηλικιωμένου, αλλά αντίθετα επιτρέπει μια μεγαλύτερη προσέγγιση ε, ηλικιωμένων και νέων και συνεργασία των γενναιών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η Μάριον Χάρκιν έχει το λόγο. Ωραία, πρώτο λοιπόν, κύριο Κοσλόφσκι, ευχαριστώ πολύ. Αναλύοντας το κείμενο το οποίο εκπώνησε η Κομισιόν αλλά και το κείμενο του συναδέλφου Κάστλε, ε, σκέφτηκα κάποια σχόλια το οποίο θέλω να σας μεταφέρω. Το πρώτο έχει να κάνει με την παράγραφο 12 και αφορά την αύξηση του αριθμού ηλικιωμένων ε, που απασχολούνται και επίσης επικέντρωση στην καινοτομία, στην καινοτομία υψηλού επίπεδου. Νομίζω ότι αυτό είναι δυνατόν, μπορεί να βοηθήσει καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες, μπορεί να βοηθήσει στην ε, υπέρβαση κάποιων προβλημάτων που σχετίζονται με την υγεία, αλλά να βοηθήσει και την επαγγελματική οργάνωση. Ίσως καλό θα ήταν να αναπτυχθούν και κάποια προσόντα ε, σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής ε, σταδιοδρομίας, αλλά να υπάρχουν ε, και οι κατάλληλες δεξιότητες για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες του πιο ηλικιωμένου πληθυσμού. Μεταφορά γνώσεων, μεταφορά εμπειρίας, κοινωνικές δεξιότητες. Σε αυτός τους τομείς μπορεί να κάνει πάρα πολλά η πιο ηλικιωμένη γενιά να μεταλαμπαδεύσει αυτές τις γνώσεις και την εμπειρία της στους νεότερους. Είπατε ότι είναι το ευρωπαϊκό έτος του εθελοντισμού το τρέχον έτος. Και ίσως κάποια θέματα από αυτό το χρόνο θα πρέπει να τα περάσουμε και στο επόμενο έτος, να προωθήσουμε δηλαδή και κάποια ε, καλά ε, παραδείγματα της συνεργασίας και της αλληλεγγύης μεταξύ των γενναιών και στον τομέα τη εθελοντική συνεργασία. Υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα τα οποία θα πρέπει να συμμετέχουν. Το ευρωπαϊκό επίπεδο, το εθνικό επίπεδο, το περιφερειακό και το τοπικό επίπεδο, αλλά βέβαια και οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Όλοι οι εταίροι πρέπει να συμμετέχουν γιατί είμαι πεπισμένο ότι όλοι έχουν να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο. Γι' αυτό το λόγο υποστηρίζω την ιδέα να έχουμε το Ευρωπαϊκό έτος 2012, έτος της ενεργού γύρανσης. Ευχαριστώ και τώρα η Μαριάν Χάρκιν. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εξαιρετική του δουλειά που περιλαμβάνει πολύ ωραίες ιδέες. Θα υποστηρίξω και αυτό που είπε ο φίλος ε, Γέλκο Κασί και κάποια άλλα σύντομα σχόλια. Νομίζω ότι κάποιοι προλαλήσαντε ήδη μίλησαν για τη σχέση μεταξύ των διαφόρων ε, ε, ετών, τη διασύνδεση όπως αυτή που θέλουμε να είναι μεταξύ του έτους αθλητισμού και του έτους ενεργογύρανσης. Είναι και τα δύο ε, στο πλαίσιο της ελληνική δράσης εξαιρετικά σημαντικά. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό τα αίτια αυτά να τα συσχετίσουμε, να τα συνδέσουμε μεταξύ του και να υπάρχει μια συνέργεια. Και βέβαια, όταν ολοκληρώνεται το ένα έτος δεν έχει τελειώσει εκεί και είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει συνέχεια. Νομίζω ότι ένας από τους τρόπους για να το εξασφαλίσουμε αυτό είναι οι ηλικιωμένοι, ε, τους χάρη κοινοβούλια ηλικιωμένων και κάποιε άλλε ομάδε να μπορούν να συμμετέχουν Παραδείγματο χάρη για το 2011 υπάρχει ένα δίκτυο 33 μη κυβερνητικών οργανώσεων που συνεργάζονται με την Κομισιόν και το Κοινοβούλιο για να εξασφαλίσουν την επιτυχία του ευρωπαϊκού αυτού έτου. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό η προσέγγιση αυτή να μην είναι από πάνω προς τα κάτω μόνο, αλλά και αντίστροφα από κάτω προ τα πάνω. Και επίση να υποστηρίξω και κάποιε από τι τροπολογίε τη Επιτροπή Ρέτζι, όπου γίνεται λόγο για την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι και οι τοπικοί και οι περιφερειακοί φορείς θα συμμετάσχουν ενεργά και θα συντονίσουν τι δράσει με τι ε, προεδρίε και με την Κομισιόν. Και ένα τελευταίο σχόλιο. Συντάξει που επανέρχεται και σε αυτή την έκθεση το θέμα, νομίζω είναι η τροπολογία 14, όπου η συγητή μιλά και πάλι για τους τρεις πυλώνες. Έχοντας ακούσει τη συζήτηση σήμερα το πρωί, δεν νομίζω να υπάρξει πλήρη συμφωνία από το σημείο αυτού, και ίσως και εγώ να καταθέσω μια τροπολογία σχετικά. Αλλά κατά τα υπόλοιπα είναι εξαιρετική έκθεση. Ευχαριστώ. Κάποια σχόλια και εγώ ήδη από το στο λόγο στον κύριο Κάσπερ. Είναι πολύ σημαντικό να συμπεριλάβουμε και τα άτομα με αναπηρίε όταν μιλάμε για την ενεργό γύρανση, γιατί πολλά άτομα βέβαια στην ηλικία αυτή έχουν προβλήματα και αναπηρίε όπω και νέοι. Στην τροπολογία 16 μιλάμε για μια θετική ε, ένα θετικό αποτέλεσμα. Αυτό το οποίο με απασχολεί εμένα είναι ότι σε όλα τα ευρωπαϊκά έτη έχουμε συνδιασκέψεις, έχουμε συναντήσεις, χτυπάμε με ευχαρίστηση τον εαυτό μας στην πλάτη, λέμε τι ωραία που τα καταφέραμε. Αλλά όταν βλέπουμε τη συνέχεια η οποία δίνεται, δεν υπάρχει συνέχεια, απλώς προχωρούμε στο επόμενο έτος. Είναι απαραίτητο λοιπόν να δώσουμε σάρκα και ωστά σε αυτέ τι πρωτοβουλίε και να μιλήσουμε περισσότερο για τα αποτελέσματα που θέλουμε να πετύχουμε. Και ένα από αυτά τα αποτελέσματα, και δεν σα εκπλήσει αυτό, είναι το να πούμε ότι η οδηγία, η οζόλια οδηγία κατά των διακρίσεων σε σχέση με την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίε, καλύπτει και τι ηλικίε βέβαια και όλα αυτά, θα πρέπει να ξεπεραστεί το μπλοκάρισμα που υπάρχει στο Συμβούλιο και να εγκριθεί. Ξέρουμε ότι έχει ε, μπλοκάρει στο Συμβούλιο Υπουργών για πάρα πολύ καιρό και θα είναι πάρα πολύ θετικό να εξασφαλίσουμε ότι θα προχωρήσει αυτή, αυτό το νομοθέτημα στο Συμβούλιο γιατί υπάρχει ένα κράτος μέλος αυτή τη στιγμή που εμποδίζει να ευδοκιμήσει αυτό το νομοθέτημα. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα εμπλακούν και οι ΜΚΟ και τα θετικά αποτελέσματα που προσδοκούμε από αυτό το έτος θα πραγματοποιηθούμε και να μπορούμε στο τέλος του χρόνου να πούμε ναι, πετύχαμε κάτι και στη συνέχεια να οικοδομήσουμε πάνω σε αυτές τις επιτυχίες και να προχωρήσουμε. Στον κύριο Κάσλε δίνω λοιπόν το λόγο πάλι για τα τελικά του σχόλια. Σας ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τις εκτιμήσεις. Άκουσα πολύ προσεκτικά τις επιθυμίες για κάποιες αλλαγές. Θα ήθελα να αναφερθώ στα κεντρικά σημεία, έτσι όπως ε, τα άκουσα. Χαίρομαι γιατί όλοι θεωρούν και συμφωνούν ότι ο τίτλος είναι κάπως σύντομος. Ευρωπαϊκό έτος ενεργούς γύρασης 2012. Θα πρέπει ε, να συμπεριλάβουμε ενδεχομένως στον τίτλο και κάτι που να αναφέρεται στην αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών έτσι ώστε να συμπεριλάβουμε και τις προτάσεις όλων όσων αναφέρθηκαν στο θέμα αυτό. Όλοι το έθιξαν αυτό το θέμα της αλληλεγγύης. Ίσως λοιπόν θα χρειαστεί ένας υπότιτλος. Πώς οι ηλικιωμένοι θα μπορέσουν να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Η αξιοπρέπεια είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο βεβαίως δεν εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από ένα επίδομα, από κάποιες αποδοχές, από ένα εισόδημα. Η αξιοπρέπεια συμπεριλαμβάνεται και σε κάποιες άλλες πτυχές. Το θέμα επίσης της ζωτικότητας. Πώς μεταφράζεται η λέξη αυτή. Βιταλιτέ. Vitality. Με ποιο τρόπο λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί θα μπορέσουν να ζήσουν με αξιοπρέπεια και με ζωτικότητα, με ενέργεια. Αυτά τα δύο στοιχεία πρέπει κάπου να τα αναφέρουμε ε, στον τίτλο ή στον υπότιτλο. Θέλω πραγματικά να εστιάσω την προσοχή μου σε αυτήν την γενιά, την οποία την ονομάζουμε Silver Generation, ασημένια γενιά αυτή τη γενιά την οποία θέλω να βοηθήσω, να βοηθήσουμε έτσι ώστε να ζήσει καλύτερα στην Ευρώπη. Έτσι ώστε να μπορέσει να δώσει και να πάρει από την κοινωνία μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και αυτό εξάλλου νομίζω ότι είναι και το κοινό σχόλιο των περισσότερων συναδέλφων. Υπάρχουν πολλές τροπολογίες και ελπίζω να μην φτάσουμε σε μια παρόμοια κατάσταση με αυτή που αντιμετωπίζουμε σήμερα με την έκθεση για τις συντάξεις, δηλαδή ένα πολύ μεγάλο αριθμό τροπολογιών που μετά πρέπει να τις επεξεργαστούμε στις συμβαστικές τροπολογίες, το θέμα δηλαδή που θα ψηφίσουμε σήμερα το απόγευμα. Τώρα, τι εννοούμε ενεργός ηλικία. Ενεργός ηλικία είναι η ηλικία που ξεκινάει με τη γέννηση ενός ανθρώπου. Από την αρχή λοιπόν θα πρέπει να ξεκινήσουμε να αντιμετωπίζουμε αυτήν την ηλικία. Πρόβλεψη και βεβαίως ευελιξία είναι δύο βασικές αρχές. Το θέμα της υγείας, το οποίο βεβαίως ξεκινάει από τη γέννηση ενός ανθρώπου μέχρι το θάνατό του. Όσον αφορά το θέμα των συντάξεων, βεβαίως αυτό είναι αντικείμενο και πολλών άλλων εκθέσεων. Ο ρόλος των μη κυβερνητικών οργανισμών που θεωρώ πολύ σημαντικούς φορείς, εταίρους ε, στην συζήτηση αυτή και θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο, όχι ίσως τον τίτλο, αλλά κάπου να τους αναφέρουμε. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική η συνεισφορά όλων των κρατικών φορέων, του ευρωπαϊκού βεβαίως επίπεδου, αλλά μέχρι το τελευταίο περιφερειακό τοπικό επίπεδο. Δεν έχει σημασία να οργανώνουμε συνέδρια και συνδιασκέψεις εδώ στις Βρυξέλλες ή στις πρωτεύουσες των κρατών μελών. Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουν ότι η ευαισθητοποίηση γίνεται σε όλα τα επίπεδα. Και νομίζω ότι εδώ μπορεί να υπάρξουν τροπολογίες. Γιατί όλα τα ευρωπαϊκά έτη που οργανώνουμε, για όλα τα θέματα, θα πρέπει να έχουν μια συνέχεια και μια συγκεκριμένη παρακολούθηση όταν τελειώσει παραδείγματο χάρη το 2012 πώς μπορούμε να παρακολουθήσουμε τις επιπτώσεις αυτής της δράσης και αυτό όχι μόνο για το 2012 και το έτος της ενεργούς ε, γύρανσης αλλά για όλα τα ευρωπαϊκά έτη. Σας ευχαριστώ. Um, Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. 11 Φεβρουαρίου είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό στις 16 Μαρτίου εδώ στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια του Μαΐου. Συγγνώμη, έκανα λάθος, λέει η πρόεδρος. 9 Φεβρουαρίου στις 12 είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Προχωρούμε στο επόμενο θέμα με την κυρία Στάινροκ. Νεολαία σε κίνηση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα όσον αφορά την βελτίωση των εκπαιδευτικών συστημάτων και την ενσωμάτωση των νέων στην αγορά εργασίας. Βελτίωση της κινητικότητας που είναι προϋπόθεση για την επιτυχία στην Ευρώπη αυτής της προσπάθειας. Σήμερα βλέπουμε ότι αυξάνεται ο αριθμός των νέων που είναι άνεργοι και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην έχουμε κανέναν νέο στην Ευρώπη στο περιθώριο. Η πρόταση της Επιτροπής Youth on the Move, νεολαία σε κίνηση, είναι ένας από τους σημαντικούς στόχους για την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020. Μέτρα κλειδιά για την αύξηση της ελκυστικότητας και τη βελτίωση των εκπαιδευτικών συστημάτων καθώς και των συστημάτων επαγγελματικής κατάρτισης στην Ευρώπη. Εδώ δεν θέλουμε απλώς να ξαναδούμε τα υπάρχοντα μέτρα και εκπαιδευτικά συστήματα, αλλά πραγματικά να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε επιπλέον. Να μην παραμείνουμε λοιπόν στις δηλώσεις, στα λόγια και στις προθέσεις. Σήμερα βλέπουμε ότι από τις προτάσεις της Επιτροπής λείπει το θέμα της χρηματοδότησης αυτής της κινητικότητας δεν αναφέρεται παραδείγματο χάρη οι ασκήσεις των νέων, τα εκπαιδευτικά προγράμματα άσκησης, επαγγελματική άσκησης, κάτι πάρα πολύ σημαντικό για νέους, ιδιαίτερα για νέους από πολύ ευάλωτε και αδύναμες κοινωνικέ ομάδες, για τους νέους ε, οι οποίοι προέρχονται από οικογένειες μεταναστών, τους Ρώμα, θέμα που αναφέρθηκε εξάλλου και στην Ολομέλεια, θα πρέπει να δούμε πολύ περισσότερο τα δικαιώματα αυτών των ομάδων. Χρειαζόμαστε κάποια ελάχιστα πρότυπα και για τις περιόδους επαγγελματικής άσκησης, αλλά και για την περαιτέρω επαγγελματική κατάρτιση το θέμα της τεχνολογίας, της καινοτομίας, πρέπει να προετοιμάσουμε τους νέους μας για τους τομείς αυτούς. Επίσης, σήμερα ξέρουμε ότι δεν είναι μόνο θέμα κοινωνικής ασφάλισης, είναι πολύ σημαντικό το θέμα της συναπόφασης. Εγώ το υπογραμμίζω αυτό, γιατί πολλές φορές βλέπουμε οι νέοι να μην έχουν καμία απολύτως προοπτική. Πρέπει επίσης να δούμε ότι η νεολαία σε κίνηση δεν μπορεί να επιτευχθεί παρά μόνο με την συμμετοχή των ίδιων των νέων. Η κινητικότητα πρέπει να είναι κάτι που το αποφασίζουν οι νέοι, πρέπει να συμβαδίζει με την προσωπική του ζωή και βεβαίως αυτή η βελτίωση της εκπαιδευτικής και επαγγελματική κατάρτισής τους θα πρέπει να αποφασιστεί σε κάποια συγκεκριμένη περίοδο της ζωή τους από τους ίδιου του νέου. Το θέμα τη ποιότητα αυτή της κατάρτιση, εκπαιδευτική και επαγγελματική είναι πολύ σημαντικό και επαναλαμβάνω, εδώ θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ιδιαίτερα το θέμα της επαγγελματικής άσκησης, που επαναλαμβάνω δεν αναφέρεται στην έκθεση αρκετά. Προσπάθησα να συγκεντρωθώ σε κάποια σημεία καθοριστικά, σημεία κλειδιά για τις τροπολογίες. Έχω πολλές ιδέες και ξέρω ότι οι τροπολογίες σίγουρα θα αποσαφηνίσουν το κείμενο δεν υπάρχουν όμως πολύ μεγάλες διαφορές θα έλεγα μεταξύ των ε, πολιτικών ομάδων. Ε, υπήρξε πολύ καλή συνεργασία με όλους ε, στην Επιτροπή και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε με πολύ επικοδομητικό τρόπο να καλύψουμε τα κάποια κενά αυτής της έκθεσης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φεράτη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να τονίσω τη σημασία της πρωτοβουλίας νεολαίας σε κίνηση. Καρπό μια συζήτηση και συνένεση για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας που είχε τεθεί ως πολιτική προτεραιότητα της Ισπανικής Προεδρίας. Με τη βοήθεια της Βελγικής και Ουγγρικής Προεδρίας ήδη βλέπουμε τα πρώτα αποτελέσματα, γίνονται τα πρώτα βήματα. Αυτή η πρωτοβουλία επιτρέπει να μπουν οι νέοι στο επίκεντρο της πολιτικής ατζέντας Ευρωπαϊκής Ένωσης ως αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος αλλά και του μέλλοντος για να οικοδομηθεί το μέλλον της Ευρώπης. Ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι το σημερινό πλαίσιο, γι' αυτό λοιπόν η προτεραιότητα να βοηθήσουμε τους νέους να έχουν τα απαραίτητα και επαρκή μέσα για να χτίσουν ένα αξιοπρεπέ μέλλον. Διότι είναι τεράστιε οι δυσκολίε που αντιμετωπίζει στον εργασιακό χώρο ένα νέο σήμερα. Πράγματι, όπω λέγεται και στην έκθεση και στην ανακοίνωση, το εκπαιδευτικό έλλειμμα των νέων έχει άμεση σχέση με, τις, ε, με τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας. Αλλά πρέπει να πω ότι ακόμη και μεταξύ των νέων σήμερα ως κοινός παρονομαστής στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει μεγάλη δυσκολία στη μετάβαση από το σύστημα, το εκπαιδευτικό στο παραγωγικό σύστημα. Δεύτερον και παρά, παρά ε, ε, των, διαφορών μεταξύ των διαφόρων κρατών υπάρχει και το χρονικό στοιχείο που είναι κοινό σε όλα τα κράτη-μέλη διότι δεν υπάρχουν ε, κάποια της περιορισμένου χρόνου συμβάσεις. Επίσης είναι δύσκολο να περάσει κανείς από συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου εργασίας. Υπάρχει επίσης και το θέμα της μερικής απασχόλησης. Κάποιες φορές εκπαίδευση ή μελέτη δύσκολα συμβαδίζει με την απασχόληση και υπάρχουν και δυσκολίες για να υπάρξουν μεγαλύτερες δεξιότητες και ικανότητες για τους νέους. Συμφωνώ επίσης και με αυτό που είπε η συγγήτριά μας, δηλαδή ότι η μείωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων δεν προωθεί την απασχολησιμότητα. Είναι ένα πρόβλημα αυτό των τελευταίων δέκα ετιών. Νομίζω ότι απο... απέτυχε Δηλαδή, παρότι είχαμε ακολουθήσει αυτή την τάση μείωση των εγγύσεων, μείωση των προνομίων, τελικά δεν μειώθηκε η διαφορά που υπάρχει μεταξύ ε, του, γενικού ποσοστού ανεργίας και του ειδικού ποσοστού της νεανικής ανεργίας. Τέλος πάντων, το ποσοστό της νεανικής ανεργίας μέσα στο γενικό ποσοστό ανεργία. Νομίζω ότι είναι και διπλάσιο. Τώρα, σε ό,τι αφορά, ε, σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε πάνω από 5 εκατομμύρια νεαρού ε, και έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει σχέση μεταξύ εγκατάλειψη του σχολείων, επαρκού εκπαίδευση και ποσοστού ανεργία. Για όλου αυτού του λόγου νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική η πρόταση να έχουμε την απλή και φιλόδοξη συνταγή τη μεγαλύτερη εκπαίδευση, για καλύτερη απασχόληση, λιγότερα γραφειοκρατικά εμπόδια. Αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο. Σήμερα ε, υποστηρίζουμε όλο και περισσότερο την ποιοτική απασχόληση που απαιτεί συγκεκριμένε δεξιότητε, γνώσει ε, και εμπειρίε. Με βάση ε, κάποιε μελέτε τη Κομισιόν, στο 95% των θέσεων εργασίων χρειάζονται υψηλέ δεξιότητε και στο 50% μέσε δεξιότητε και επίση και θεωρείται πολιτιστική, οι πολιτιστικέ γνώσει, η γλωσσομάθεια κτλ. Πρέπει λοιπόν να ε, βοηθήσουμε τη στρατηγική αυτή πρέπει να καταπολεμήσουμε την πρόρη εγκατάλειψη του σχολείου. Και σε αυτό το ευρωπαϊκό πλαίσιο νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε την ανταλλαγή καλύτερων πρακτικών και να αξιοποιήσουμε τη συνεργασία μεταξύ κομισιών και διαφόρων ιδρυμάτων και πανεπιστημίων σε, στα κράτη-μέλη. Θα ήθελα να κάνω και κάποια συγκεκριμένη πρόταση, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι σε κάθε σύμβαση προβλέπονται τα ευρεία και αξιοπρεπή δικαιώματα. Θα πρέπει να υπάρχουν και κάποιες ελάχιστες κατευθυντήριες γραμμές, πιστεύω, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως ένας κατάλογος των ελάχιστων ε, ε, δικαιωμάτων των ε, νεαρών εργαζομένων. Παραδείγματο χάρη, περίοδοι άσκηση, υποτροφίε ή ε, η κατάσταση γενικά που έχουμε στις υποτροφίες, στους υποτρόφους, στα διάφορα κρατημέρια, γιατί υπάρχουν διαφορές. Πρέπει να υπάρξει κάποια ελάχιστα εναρμόνιση. Επίσης είναι πολύ ε, σημαντικό ε, τα κοινωνικά ταμεία, τα κονδύλια του κοινωνικού ταμείου να προορίζονται σε μεγάλο βαθμό και για την ενική απασχόληση δεδομένων των εθνικών δυσκολιών. Πρέπει λοιπόν κατά προτίμηση και κατά προτεραιότητα να δίνονται εκεί κάποια κονδύλια και θα πρέπει επίσης και στην έρευνα να δώσουμε έμφαση. Έχουμε την οικονομική κρίση, η οποία έδειξε πόσο σημαντικό είναι το, όργανο, το εργαλείο των επενδύσεων. Πρέπει λοιπόν να υπάρξουν επενδύσει. Θα πρέπει να γίνουν μεγαλύτερε διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει σε κοινοτικό επίπεδο. Οι Γενικέ γραμμέ, όπω είπα, συμφωνώ με την απόψη την οποία μας παρουσίασε η σύντροφος Γιώτα και νομίζω ότι μπορούμε να επεξεργαστούμε την τελική έκθεση στον ένα στο δυνατόν πληρέστερ γιατί όπως είπα η νεολαία σε κίνηση είναι κάτι που αν το δούμε με επαρκή φιλοδοξία, νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε ε, πολύ ελπίδα στα εκατομμύρια των νέων που προσβλέπουν σε αυτό. Ευχαριστώ. Thank you. Ε, ευχαριστώ. Ο Ζώος και μετά η Μάριο Χάρκιν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λέει κύριος Μπαχ. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Στάινρουκ για αυτά που είπε. Είναι μια πολύ σημαντική συνεισφορά στην γενική προβληματική και εγώ συμφωνώ απόλυτα με τον Λίσαντα, Είναι, είναι προφανώς το μέλλον της Ευρώπης. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα που έχει καταστροφικές διαστάσεις. Μιλάνε όλοι για μια χαμένη, μιλάνε πολύ για μια χαμένη γενιά, επομένως πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που είναι στη διάθεσή μας για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα και νομίζω ότι με αυτή την γνωμοδότηση δίνουμε μια σημαντική συμβολή στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Έχουμε το πρόβλημα με το άρθρο 50 του κανονισμού. Είμαστε συνδεόμενοι επιτροπή βέβαια καταρχήν. Τίθεται το θέμα της, ε, των αρμοδιοτήτων επίσης, το θέμα της επικουρικότητος, για την κατάρτιση και την εκπαίδευση φυσικά σε μεγάλο βαθμό εναπόκειται στις αρμοδιότητες των κρατών μελών. Παρ' όλα αυτά μπορούμε εμείς να συμβάλλουμε σημαντικά. Επειδή έχει προχωρήσει και ο χρόνος, θα κάνω μονάχα μερικέ σύντομες παρατηρήσεις στα υπόλοιπα σημεία και κάποια ερωτήματα στο σημείο 2. σε ό,τι αφορά τα, το μη περιορισμό των κοινωνικών δικαιωμάτων μέσω των ε, συμβάσεων εργασίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να επιληθεί σε επίπεδο κρατών μελών. Για το σημείο 3, την πρωτοβουλία για τους δείκτες σε ό,τι αφορά τις ομάδες ε, στόχων, εδώ φοβάμαι ότι ίσως ε, δημιουργούμε ένα πρόσθετο στατιστικό άγχος και είναι πάρα πολλές οι πολιτικές οι οποίες κατευθύνονται μονάχα από στατιστικά στοιχεία ενώ αυτές οι στατιστικές πολλές φορές ε, δεν είναι πλήρεις και βασίζονται σε διαφορετικές ε, προσεγγίσεις και έχω κάποιες ε, αμφιβολίες σε σχέση με το πρόσφορο μιας τέτοιας προσέγγισης. Επίσης το θέμα των προσόντων, η επίσημη αναγνώριση των προσόντων και αυτό θα μπορούσε να είναι πρόβλημα. Έχουμε δει ήδη πολλές δυσκολίες να υπάρχουν για την αμοιβαία αναγνώριση των προσόντων μέσα στα κράτη-μέλη, μεταξύ των κρατών μελών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εμείς θα πρέπει να εξασφαλίσουμε σαφήνεια και όχι περαιτέρω δυσκολίες. Και επίσης τα κρατικά επιδοτούμενα προγράμματα για την εργασία των νέων. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν τέτοια προγράμματα σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εδώ θα πρέπει να ακολουθήσουμε το υπόδειγμα των βελτίστων πρακτικών για να μπορέσουμε να μεταλαμπαδεύσουμε αυτές τις εμπειρίες για τις ε, συμβάσεις περιορισμένου χρόνου. Αυτό μου φαίνεται ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει. Ότι οι νέοι με τον τρόπο αυτό, με τις ε, ε συμβάσεις αυτές περιορισμένου χρόνου, απενάντως από τη μία σύμβαση στην άλλη, δεν μπορούν να οικοδομήσουν μια ε, μια καριέρα. Δεν ξέρω λοιπόν πώς θα μπορούσε να υπάρχει μια σωστή πολιτική σε φορολογικό επίπεδο στις φορολογία της εργασίας που να προωθεί τι συμβάσει αορίστου χρόνου. Αυτό όμως παραμένει μέσα στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, η φορολογική πολιτική όπως γνωρίζουμε όλοι. Εμείς θέλουμε επίσης να έχουμε δημόσιες διοικήσεις οι οποίες λειτουργούν καλύτερα. Εγώ έχω δει σε πολλά κρατημέλη μόνο 5-10% των νέων να παίρνουν θέσεις εργασίας μέσω των δημοσίων μηχανισμών εξέβρεσης εργασίας και ίσως θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι δημόσιες διοικήσεις και οι δημόσιοι φορείς θα παίζουν ένα σημαντικότερο ρόλο. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ για τη συνεργασία που υπήρξε μεταξύ μας. Νομίζω ότι αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική γνωμοδότηση και ένα έγγραφο το οποίο έχει μεγάλη αξία. Ευχαριστώ. Uh, uh Η Μάριον, σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω και εγώ την εισηγήτρια για τη γνωμοδότησή της. Η σκιώδη μας εισηγήτρια είναι αδιαχείριση, είναι σε μια άλλη επιτροπή και ψηφίζει και γι' αυτό μου ζήτησε να κάνω εγώ τα σχόλια εξ ονοματός και θα προσθέσω και ορισμένα δικά μου. Η Νάντια υποστηρίζει την άποψή σα για την κινητικότητα των νέων και τη σημασία τη κινητικότητα. αυτής. Χαίρομαι πάρα πολύ που στην παράγραφο 4 έχετε μια <clears throat> φράση που αναφέρεται στην κινητικότητα για το στόχο τη απασχόληση. Γιατί μερικέ φορέ όταν μιλάμε για κινητικότητα είναι σαν να είναι απλώς μια γενική κινητικότητα. Δεν πρόκειται εδώ για εκπαίδευση ή κατάρτιση ή ακόμα και για τουρισμό, αλλά για απασχόληση. Υποστηρίζει επίσης συνάντια την πρωτοβουλία EURES που αναφέρεται στο αρχικό σχέδιο και τονίζει ότι πρέπει να μειωθεί ο αριθμό αυτών που δεν τελειώνει το σχολείο. Επίσης έχουμε το σχόλιο στην παράγραφο 2 που ανέφερε και ο προηγούμενος ομιλητής, τον περιορισμό των κοινωνικών δικαιωμάτων. Είπε ότι εκεί μπορεί να υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να μην εμποδίσουμε τους νέους να αποκτήσουν μια πρώτη θέση εργασίας. Και τα δικά μου τώρα σχόλια πέραν της Ναδίας είναι ότι συμφωνώ πάρα πολύ με την παραγραφό 3 όπου αναφέρεται ότι η πρόοδος θα πρέπει να παρακολουθείται καθ' όλη τη διάρκεια της εφαρμογής αυτών των προγραμμάτων και θα πρέπει να γίνεται αυτή η παρακολούθηση μέσα από μια σειρά ενδεικτών και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Θα είναι πολύ σημαντικό από τη δική μας πλευρά να εξασφαλίσουμε τη στρατηγική της Ευρώπης 2020 επιτυγχάνει τους στόχους της. Ξέρω ότι η γνωμοδότηση είναι μέσα σε ένα πλαίσιο βελτίωση του συστήματο εκπαίδευση και κατάρτιση Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σημαντικό να συνδέσουμε την εκπαίδευση και την κατάρτιση με τι θέσει απασχόληση δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε τη μακροοικονομική κατάσταση η οποία υπάρχει στα κράτη-μέλη, δεν λειτουργούμε σε κενό αέρος και ίσως θα μπορούσαμε με κάποια τροπολογία να προσθέσουμε και αυτή τη μνήα της μακροοικονομικής κατάστασης, του γενικού πλαισίου στο οποίο βρισκόμαστε. Τελικό σχόλιο στην παράγραφο 10. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με την συγγήτρια όταν λέει ότι χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις μαθητείες. Και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό να έχουμε ένα σωστό ευρωπαϊκό υπότιμο για αυτές τις διαδικασίες. Η κυρία Στάιν Ρουκ για να κλείσει. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ για όλους όσους πήραν το λόγο και έκαναν κάποιες παρατηρήσεις και υποδείξεις. Χαμένη γενιά. Ναι, χαμένη γενιά ε, εκ των οποίων πολλοί θα έπρεπε σήμερα να βρίσκονται στην αγορά εργασίας και να έχουν και μια σημαντική συνεισφορά. Στη Γερμανία το βλέπουμε αυτό καθημερινά πόσα χαμένα ταλέντα λείπουν από την αγορά. Παρ' όλα αυτά πρέπει να πω ότι γίνονται προσπάθειες έτσι ώστε να επαναφέρουμε τους νέους αυτούς στην αγορά μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, επαγγελματικών προγραμμάτων κατάρτισης σε συνεργασία με πιο ηλικιωμένους εργαζόμενους. Γι' αυτό και εδώ θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω ε, τους ε, ειδικού και εμπειρογνώμονες από το Διεθνές Γραφείο Εργασίας οι οποίοι έχουν αποδείξει ότι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ της παραμονής των ηλικιωμένων στην αγορά εργασίας και των νέων που μπαίνουν. Υπάρχουν ε, επίσης προσπάθειες για την αναγνώριση των ε, δεξιοτήτων και των προσόντων. Αυτό πολύ το ανέφεραν εχθές. Διάβασα στον τύπο, σε μια γερμανική εφημερίδα, ότι θέλει η κυρία Μέρκελ να υπάρξει ένα σύστημα αμοιβές αναγνώρισης στην Ευρώπη των δεξιοτήτων και προσόντων που να μην ξεπερνά τους 12 μήνες. Αλλά ακόμα και 12 μήνες είναι πολύ μεγάλη χρονική περίοδο. Ακόμα πιο γρήγορα θα πρέπει να γίνεται αυτή η αναγνώριση. Σήμερα βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά διαφορετικά συστήματα στην Ευρώπη. Βλέπω επίσης και τις προτάσεις σας για την αύξηση των προγραμμάτων που προσφέρονται στους νέους. Υπάρχει μια πρόταση για 10%. Αυτό είναι αρκετό. Μείωση της γραφειοκρατίας, βεβαίως, αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε όμως πιο συγκεκριμένα. Τι εννοείται μείωση της γραφειοκρατίας, για να είμαστε πιο ρεαλιστικοί. Κατά τα άλλα, συμφωνώ όσον αφορά τις αρμοδιότητες, πολλά από κοινού κάνουμε με την Επιτροπή Πολιτισμού, έτσι ώστε να βρεθούν κάποιες κοινέ προτάσεις. Ευχαριστώ. Η προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών είναι η 15η Μαρτίου, 16 θα ψηφίσουμε εδώ, τον Απρίλιο στην Επιτροπή Πολιτισμού και το Μάιο στην Ολομέλεια. Το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορά την καινοτομία μεταμόρφωση της Ευρώπης για έναν κόσμο μετά την κρίση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Ένωση Καινοτομίας είναι μια εμβληματική πρωτοβουλία με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης ε, για τη χρηματοδότηση για έρευνα και καινοτομία, ώστε καινοτόμε ιδέε να μπορούν να δημιουργηθούν προϊόντα και υπηρεσίε που θα δημιουργούν με τη σειρά του ε, ανάπτυξη και απασχόληση. Όλα αυτά βέβαια είναι πάντοτε σημαντικά, ιδίω όμω σήμερα με την συνεχιζόμενη χρηματοπιστωτική κρίση. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε πολλά στον τίτλο αυτό Ένωση Καινοτομία, αλλά στην Επιτροπή μα νομίζω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε σε ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την απασχόληση και τι κοινωνικέ υποθέσει. Και πράγματι, θα πρέπει η έρευνα και η καινοτομία να διαδραματίσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο για την οικονομική ευημερία και για την αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων. Η καινοτομία θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να αντιμετωπιστούν σημαντικέ προκλήσει στην Ευρώπη, όπω δημογραφικέ αλλαγέ, σημαντικά προβλήματα στον τομέα τη υγεία, κοινωνικά προβλήματα και γι' αυτό κατά τη, νο... κατά γνώμη πρέπει να τονιστεί η σημασία των συμπραξιών ιδιωτικού δημόσιου τομέα. Θα ήθελα επίσης να συστήσω να εκμεταλλευτούμε εκμεταλλευτούμε τις ε, δυνατότητες ε, δημιουργίας εταιρικών σχέσεων που σε κάποια κράτη-μέλη γίνεται πιο γρήγορα από ό,τι σε κάποια άλλη. Χρειαζόμαστε αυτές τις πιλωτικές ε, συμπράξεις εταιρικές σχέσεις και περιμένω να δρομολογηθούν και άλλες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κοινωνική καινοτομία θα μπορούσε να αποτελέσει και κεντρική προτεραιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και των προγραμμάτων του. Για να ενισχυθεί η καινοτομία στην κοινωνία χρειάζεται διαβίου μάθηση, χρειάζονται μεγαλύτερα εκπαιδευτικά επίπεδα και περισσότερη κατάρτιση για όλες τις ηλικιακές ομάδες. Ιδίως ε, η καινοτομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επικεντρώνεται σε τομείς που γεννούν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη. Κοινωνία, ε, ε, τεχνολογίες πληροφοριών ε, και επικοινωνιών, ε, πάνω από 700 δις, πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη παράγεται από αυτό το τομέα. Οι ικανότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα TPE... είναι κάτι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να ευνοηθεί η χρήση των ανοιχτών κωδίκων και άλλων τέτοιων μεθόδων και πρέπει να βοηθηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι πολίτες ώστε να συμμετάσχουν σε αυτές τις αναπτυξιακές διαδικασίες, ε, διαδικασίες ανάπτυξης νέων υπηρεσιών. Ένα τελευταίο ζήτημα το οποίο θέλω να αναφέρω είναι ότι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Καινοτομία θα πρέπει να εναρμονιστεί για να υπάρχει καλύτερη διακυβέρνηση, πιο εύκολη πρόσβαση ε, στη χρηματοδότηση και μικρότερη γραφειοκρατία, αλλά και για να είναι πιο εστιασμένη. Και γι' αυτό θα πρέπει να δημιουργηθεί ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας και θα πρέπει οι ερευνητές να βοηθηθούν ώστε να μπορούν να μετακινούνται ελεύθερα από χώρα σε χώρα χωρίς εμπόδια. Θα πρέπει επίσης να προωθήσουμε και ε, επενδύσεις ε, σε κεφάλαιο, με κεφάλαιο επιχειρηματικού κινδύνου σε επιχειρήσεις που έχουν το μεγαλύτερο δυναμικό. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία θα ήθελα να αναφέρω και τώρα είμαι έτοιμη να ακούσω τις δικές σας απόψεις. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Η Edith Ιστρέλα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να υπογραμμίσουμε τη σημασία του ζητήματος αυτού και θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια για την προσέγγιση της. Η καινοτομία είναι η βάση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για, τα, για το 2020 και περιέχει ένα τεράστιο δυναμικό όπως έχει δεχτεί για την δημιουργία θέσεων απασχόλησης και συγχρόνως συμβάλλει στην αντιμετώπιση της δημογραφικής γύρανσης των προβλημάτων που προκύπτουν για, το, για τα συστήματα υγείας, των αρνητικών αποτελεσμάτων της κλιματικής αλλαγής κτλ. Επομένως η καινοτομία θα πρέπει να οδηγήσει σε μεγαλύτερη συνέργεια και να δημιουργήσει πράσινες θέσεις εργασίας και, και να μπορέσει να αντιμετωπίσει στόχους ανάπτυξης που είναι ευφυής, περιεκτική και καινοτόμη προς όφελος της Ευρωπαϊκής Στατικής 2020. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι θα είναι δυνατόν να δημιουργηθούν 3 εκατομμύρια να δημιουργηθούν ε, εκατομμύρια θέσεις εργασίας και επίσης να χρησιμοποιηθούν 800 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2025. Ο στόχος επίσης είναι μέχρι το 2020 να δίδεται το 3% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην έρευνα και την ανάπτυξη. Έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να έχει και στον τομέα της, ε, των, της έρευνας και της ανάπτυξης ένα εκατομμύριο παραπάνω θέσεις εργασίας με μεγαλύτερη συμμετοχή και των γυναικών. Μας λείπουν οι γυναίκε στον τομέα τη έρευνα και τη ανάπτυξη πρέπει να αναπτύξουμε περισσότερες τέτοιε θέσει εργασία. Πρέπει εξάλλου να ενισχύσουμε τη συνεργασία μεταξύ της ε, ανώτατης εκπαίδευση και του επιχειρήν. Να έχουμε μεγαλύτερη συνέργεια και να έχουμε καλύτερα έτσι αποτελέσματα. Για όλου αυτού τους λόγους θεωρούμε επιθυμητό ότι παρά την κρίση και τα μέτρα λιτότητος, τα κράτη-μέλη δεν πρέπει να μειώσουν την επένδυσή τους στην έρευνα και την ανάπτυξη, γιατί με τον τρόπο αυτό θα υπέσκαπτον το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το μέλλον του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αυτή την εβδομάδα θα πρέπει να συζητήσει ακριβώς τα προβλήματα της ενέργειας και της καινοτομίας με στόχο να ενισχύσει τη συνειδητοποίηση της σημασίας των θεμάτων αυτών. Συμφωνούμε λοιπόν με την γραμμή που ακολούθησε η συγγήτρια. Θα επιφυλαχθούμε όμως να παρουσιάσουμε ορισμένες τροπολογίες στην γνωμοδότηση αυτή της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Επιθυμεί κάποιος άλλος συνάδελφος να παρέμβει. Ένα ερώτημα έχω εγώ, το οποίο αφορά την παράγραφο 6, ότι η καινοτομία θα πρέπει να προωθείται και μέσω κοινών διασυνοριακών ε, σχεδίων. Στην πράξη πώς το αντιλαμβάνεστε αυτό. Θα μπορούσατε να μας δώσετε κάποιες εξηγήσεις. Όχι ότι είμαι αντίθετη, δεν καταλαβαίνω ακριβώς. Τι εννοείται και πώς αυτό θα μπορούσε να δουλέψει στην πράξη. Κύριε Σαγιά, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και για τα σχόλια. Είπα ότι θα πρέπει καινοτομία, κυρία Πρόεδρε, να προωθείτε μέσω κοινών δυνασυνοριακών σχεδίων δημόσιου τομέα. Αυτό ήταν και το ερώτημά σας. Ακούστε, αυτό το οποίο λέω συγχυτίζεται με αυτό που λέει στην παράγραφο 5, δηλαδή να έχουμε έναν κοινό ευρωπαϊκό χώρο έρευνας. Και όταν μιλάμε για αυτά τα έργα ή σχέδια στο δημόσιο τομέα, πιστεύω ότι θα πρέπει ακριβώς κάτω από αυτό το τίτλο να τα εντάξουμε. Κοινά διασυνοριακά σχέδια, δηλαδή στο πλαίσιο του κοινού ευρωπαϊκού χώρου. Ευχαριστώ. Κάποιος άλλο θα ήθελε το λόγο. Όχι. Προθεσμία κατάθεση ε, τροπολογιών 11 Φεβρουαρίου. Συζήτηση των τροπολογιών 15 Μαρτίου 16 έγκριση στην Επιτροπή μας και στην Επιτροπή Ήτρε 12 Απριλίου και υπολογίζουμε στην Ολομέλεια το Μάιο. Και έτσι περνάμε στο επόμενο θέμα διαχείριση αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων νομίζω εκπροσωπεί, αντικαθιστά μάλλον την κυρία Λάμπερτ, ε, κυρία Κορνέλισεν. Ναι, πράγματι δεν μπορεί να είναι εδώ η Τζιν Λάμπερτ. Είναι η εισηγήτρια συγχρόνως και στην Επιτροπή Δημοσίου Ελευθεριών και μου ζήτησε να μπω στα παπούτσια της, θα κάνω μερικά μονάχα σχόλια και θα ακούσω μεγάλη προσοχή αυτά που έχετε να πείτε και θα τα μεταφέρω. Πρώτα απ' όλα θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι παρά τον τίτλο της ε, έκθεσης δεν πρόκειται για συζήτηση για την πυρηνική ενέργεια και αν μα αρέσει ή αν δεν μα αρέσει. Ορισμένοι βλέπουν πυρηνική ενέργεια, βλέπουν μια πράσινη εισηγήτρια και τους ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι και βγάζουν και Όχι δεν είναι θέμα πυρηνικής ενέργειας, είναι θέμα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων. Εδώ υπάρχουν ορισμένα σημεία τα οποία θέλω να θίξω. Πρώτα απ' όλα, η Τζιν θεωρεί ότι η λειτουργία, η συνδίκη μάλλον για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 153 είναι μια πιο πρόσφορη νομική βάση γιατί εδώ εμπλέκεται και η διαβούλευση με τους εργαζομένους σε θέματα υγείας και ασφάλειας. Δεύτερον, η εμβέλεια της ε, οδηγίας θα πρέπει να περιλάβει όλους τους εργαζόμενους με ραδιενεργά αναλωμένα καύσιμα. Επίσης πρέπει να υπάρχει ένας πιο περιεκτικός ορισμός των ραδιενεργών καυσίμων και των αναλωμένων καυσίμων και πρέπει να συμπεριληφθούν και τα ιστορικής προέλευσης καύσιμα στην οδηγία αυτή. Όταν αναφέρεται επίσης η εποπτεία και η επιθεώρηση από ανεξάρτητους φορείς, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, διότι ξέρουμε πόσο ολέθρια είναι τα αποτελέσματα των ανθρωπίνων σφαλμάτων. Επίσης, όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να καταλάβουν τους ενδεχόμενους κινδύνους και να είναι πλήρως πληροφορημένοι όταν εργάζονται στον τομέα αυτό. Είναι πολύ σημαντικό επίσης <clears throat> οι υπεργολάβοι να ακολουθούν αυστηρά κριτήρια για την εκπαίδευση και την ασφάλεια και να έχουν την πλήρη εμπειρογνωμοσύνη για να φέρουν σε πέρα στο έργο τους. Η πρόταση λοιπόν της εισηγήτριας περιλαμβάνει και το θέμα της ε, ε, αστικής ευθύνης για τις συνθήκες εργασίας σε μακροχρόνιο επίπεδο και πρέπει να τονίσουμε ότι δεν τίθεται το θέμα της πυρηνικής ενέργειας. Δεν συζητάμε για τα θέματα πυρηνικής ενέργειας στην Επιτροπή Απασχόλησης. Θέλουμε απλώς να εξασφαλίσουμε ότι αυτοί οι οποίοι ε, διαχειρίζονται τα πυρηνικά απόβλητα θα καλύπτονται από τις ρυθμίσεις για υγεία και ασφάλεια που, έχουν να, που πρέπει να καλύπτει όλους τους εργαζόμενους. Κυρία Στάινρουκ και μετά κυρία Μάισνερ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε με μία πρώτη εξέταση θεωρώ ότι η έκθεση της Jean Lambert είναι πλήρης, αντιμετωπίζει πλήρως τα θέματα αυτά και χρειάζεται και για μένα να υπάρξει μια διεύνηση της νομικής βάσης, να αναφερθούμε και στην χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων, τα άρθρα 114 και 115 επίσης και είναι απαραίτητο να έχουμε μια ευρύτερη σφαίρα εφαρμογής και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και για τις τροπολογίες της Jean Lambert, εγώ νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε για προστασία και θωράκιση των εργαζομένων με διάφορα συστήματα όπως είναι αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με τη ακτινοβολίες... την παρακολούθηση της υγείας των εργαζομένων και η τροπολογία 35 αναφέρεται στην αναγνώριση των ασθενειών που μπορούν να επισυμβούν στη συνέχεια ως επαγγελματικών ασθενειών με δυνατότητα έγερσης ε, αντιστοίχων απαιτήσεων εναντί των εργοδοτών. Το θέμα του ελέγχου επίσης από ανεξάρτητους φορείς είναι κάτι το οποίο έχει αναφερθεί και αυτό το οποίο εγώ πιστεύω ότι πρέπει να συμπεριληφθεί στην έκθεση είναι πιο συγκεκριμένες κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων αυτών αυτό είναι πάντα προς το συμφέρον όλων αυτών που εργάζονται με αναλωμένα καύσιμα. Νομίζω ότι η συζήτηση δεν πρέπει να περιστραφεί γύρω από το θέμα ναι ή όχι στην πυρηνική ενέργεια, αλλά να δούμε και ποια είναι η κατάσταση των εργαζομένων με τέτοια υλικά, ώστε να μπορούν και αυτοί να έχουν την απαραίτητη προστασία από την ε, ραδιενέργεια. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Τζιν Λάμπερτ. Δεν είναι βέβαια εδώ, αλλά Καταλαβαίνω για ποιο λόγο δεν είναι εδώ. Είναι ένα θέμα που φυσικά είναι αντικείμενο σοβαρής κριτικής, όχι μόνο από τους πράσινους, αλλά και από άλλους. Και αυτές όλες οι παρατηρήσεις περιγράφονται στην γνωμοδότησή της. Το θέμα των πυρηνικών αποβλήτων και των ε, χρησιμοποιημένων καυσίμων είναι ένα θέμα το οποίο το περιγράφει με πάρα πολύ ολοκληρωμένο τρόπο η συγγήτρια. Συγκεκριμένα, τι μπορούμε να κάνουμε. Εγώ πιστεύω ότι εδώ υπάρχουν τροπολογίες και παρατηρήσεις που πρέπει να υποβληθούν ακόμα. Το θέμα του σε ποιο βαθμό λεπτομέρειας πρέπει να μπούμε. Υπάρχουν ήδη ρυθμίσεις και κανονισμοί. Το θέμα είναι να δούμε τι παρακολούθηση υπάρχει. Σε γενικές γραμμές πάντως θεωρώ ότι η γνωμοδότηση είναι ε, καλή, λαμβάνονται υπόψη τα θέματα των εργαζομένων, το θέμα της προστασίας των δικαιωμάτων. Όλα αυτά περιγράφονται με ισορροπημένο τρόπο και θεωρώ ότι μπορούμε να δεχτούμε την πρόταση. Ευχαριστώ. Η ε, κυρία Εσάη, έχω μοναχά ένα ερώτημα. Αυτή η γνωμοδότηση έχει να κάνει με την ασφάλεια στον χώρο εργασία. Αυτό είναι πολύ θετικό. Το ερώτημά μου είναι το εξή όμω. Τα αναλωμένα καύσιμα και τα απόβλητα. Μήπω ε, εδώ θα πρέπει να υπάρχει και το θέμα της ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών ή όχι. Ίσως η συγγήτρια μπορεί να μου απαντήσει είναι σημαντικό να μην κινούνται αυτά τα αγαθά μέσα σε εισαγωγικά από μια χώρα σε μια άλλη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρωτού ζητήσω να λάβει το λόγο η Κομισιόν, θέλω και εγώ να κάνω κάποιε παρατηρήσει η ίδια. Νομίζω ότι είναι θαυμάσια η έκθεση τη κυρία Λάμπερτ για τις τροπολογίες 7 και 20 σε σχέση με την ανάγκη της προστασίας των εργαζομένων ανεξάρτητα από το καθεστώς ή την δραστηριότητά τους. Το θέμα είναι πώς θα καλύπτονται. Γιατί θα είναι διαφορετικοί οι κανόνες για τους εργαζόμενους που μεταφέρουν πυρηνικά, απόλυτα, απόβλητα που θα πρέπει να έχουν ιδιαίτερη προστασία. Αλλά υπάρχουν άλλοι εργαζόμενοι οι οποίοι εκτίθενται μέσα στο χώρο εργασίας θα πρέπει να καλύπτονται περισσότερο και να έχουν και περισσότερους κανόνες και οδηγίες ε, σε σχέση με την προστασία αυτή. Αυτό είναι μια διευκρίνηση λοιπόν για τις τροπολογίες 7 και 20. Και τώρα είναι το λόγο στον κύριο Χέλντον από την Κομισιόν. Καλημέρα σε όλες και όλους και σας ευχαριστώ για τις προσπάθειες που έχετε επενδύσει όλοι σε αυτό το θέμα. Επιτρέψατε μου να σας δώσω κάποιες ε, διευκρινήσεις από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την γνωμοδότηση και τις προτάσεις. Η Επιτροπή είναι πεπισμένη ότι ότι η συνθήκη Euratom ως ειδικός νόμος λέξη σπεσιάλης είναι μια καλή, ένα καλό νομοθέτημα. Ε, το άρθρο 30 καλύπτει την προστασία των εργαζομένων, αλλά έχουμε και την δευτερογενή νομοθεσία, η οποία προβλέπει την προστασία του εργαζομένου και του κοινού. Και όταν μιλάμε για δευτερογενή νομοθεσία, το κεντρικό νομοθέτημα εδώ είναι τα λεγόμενα βασικά πρότυπα υγείας. Είχαμε την οδηγία που ανατολήθηκε για τελευταία φορά το 1996 και υπάρχουν πολλά άρθρα που αναφέρονται στην προστασία των εργαζομένων αλλά και την προστασία του κοινού. Έχει να κάνει με εκπαίδευση, έχει να κάνει με όρια. Επομένως, κατά τη σύνταξη της οδηγίας εμείς έπρεπε να προσέξουμε να μην κάνουμε αλληλοεπικάλυψη με την υφιστάμενη νομοθεσία. Αυτό ισχύει και για τα βασικά πρότυπα ασφαλείας. Τώρα, όπως ε, γνωρίζετε, υπάρχει οδηγία για την ε, πυρηνική ασφάλεια, η οποία εγκρίθηκε το 2009 με την ίδια ε, βάση τη νομική, άρθρα 31-32 συνθήκης Ευρατών και βέβαια πρέπει να εξασφαλίσουμε μία συμμετρία μεταξύ των δύο οδηγιών. Πιστεύουμε λοιπόν ότι η συνθήκη Ευρατόμ είναι μια καλή βάση. Υπήρχε απόφαση δικαστηρίου μάλιστα του δικαστηρίου, οποία λέει ότι όταν έχεις ένα βασικό ζήτημα θα πρέπει να έχεις την ίδια νομική βάση. Η συνθήκη λοιπόν Ευρατόμ είναι κατάλληλη ε, βάση. Η σχετική νομοθεσία λοιπόν καλύπτει επαρκώς τους εργαζομένους ε, σε αρκετά ευρύ βαθμό και πρέπει να δούμε και τα βασικά πρότυπα ασφαλείας για να καταλάβουμε ακριβώς ε, που, ε, ότι καλύπτονται ουσιαστικά ε, τα σημεία τα οποία σας προκαλούν ανησυχία. Φυσικά είμαστε ανοιχτοί για οποιαδήποτε περαιτέρω συζήτηση του θέματος και θέλω να σας ευχαριστήσω εδώ κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Κορνέλη, τώρα ξανά το λόγο για να συνοψίσει. Ευχαριστώ. Ναι, διάφορα θέματα θίξατε. Φαντάζομαι ότι η Τζιν Λάμπερ θα μπορούσε να σας απαντήσει σε όλα και ότι θα συμπεριλάβει κάποιες από τις παρατηρήσεις σας. Θα είναι πολύ ανοιχτή φαντάζομαι όσον αφορά την νομική βάση και θα το συζητήσουμε με την Επιτροπή. Ευχαριστώ λέει Πρόεδρος. Τελειώσαμε με την ημερήσια διάταξη του πρωινού. Δεν είναι παρόντες οι εισηγητές ε, για τα υπόλοιπα θέματα και θα συνεχίσουμε το απόγευμα στις 3. Θα είμαι πάρα πολύ ακριβής όσον αφορά την ώρα έναρξης. Σας ευχαριστώ.